Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ναι. καλησπερίζω. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δεχθείτε την ημερήσια διάταξη. Μία ανακοίνωση θα κάνω μόνο, απλά να σας υπενθυμίσω From 430 to 630 Θα έχουμε λοιπόν μια συνάντηση αύριο μέχρι τις 6.30 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα αλλάξουμε τις, ε, τις, τα καρτελάκια και τις καρέκλες στην κοινή συνεδρίαση την οποία θα κάνουμε με την Επιτροπή Απασχόλησης του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Νουή, την κυρία Ντανιέλ Λουή της Εποπτικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας, για την πρώτη τακτική συνάντηση του 2016 στα πλαίσια της διοργανικής μας συμφωνίας. Φυσικά και δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται η κυρία Νουή στο Κοινοβούλιο. Είχαμε πάντα συνεχείς και καρποφόρες σχέσεις και συναντήσεις και συζητήσεις, τις οποίες εκτιμούμε δεόντως. Πάντως είναι η πρώτη τακτική μας ακρόαση και όπως όλοι γνωρίζετε υπάρχουν ε, σημαντικές εποπτικές πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε τα θέματα λοιπόν τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα λεγόμενα option and discretion. Αυτά είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποια επιπλέον θέματα τα οποία θα τεθούν ή έχουν ήδη τεθεί σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εδώ θα μας ενημερώσει η κυρία Νουή. Υπάρχουν επίσης τα συνεχιζόμενα stress και ο συγχρονισμός των διαφόρων διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, επικαλύψεις, υπάρχουν και τα λεγόμενα μεθοδολογικά θέματα, υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με τις ε, διευκρινήσεις οι οποίες έχουν γίνει για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Νομίζω ότι έχουμε και εδώ ίσως να σταθούμε λίγο, να πούμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε επίσης ε, και τα λεγόμενα ε, non-performing loans. Ε, make reference to Τα λεγόμενα κόκκινα λοιπόν δάνεια. Αυτά έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία των πιστοτικών ιδρυμάτων, έχουν σχέση με την έκθεση σε κίνδυνο των πιστοτικών ιδρυμάτων, έχουν σχέση με τη βασιλεία και γενικά είναι θέματα στα οποία θα θέλαμε να ενημερωθούμε, να εμπλακούμε και όχι απλά να κρίνουμε την εφαρμογή τους εκ των υστέρων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και γι' αυτό θα σας δώσω αμέσως το λόγο κύριε Νουή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, είναι χαρά μου που επανέρχομαι σήμερα για να αναφερθώ για την εποπτική μας εργασία. Έχουμε κάνει πρόοδο στον τομέα της αποδοτικότητας όπως επίσης και της αντοχής αλλά απαιτούνται ακόμα βήματα προόδου για την αντιμετώπιση των κινδύνων του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις θα αναφερθώ στις βασικές εξελίξεις των τελευταίο χρόνων θα επανέλθω στα θέματα της, της διαδικασίας αξιολόγησης ε, για το 2016, όπως επίσης και τα λεγόμενα National Discretions στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Νομοθεσία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με κάποιες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα ε, και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα το θέμα του ύψους και του λόγου των κεφαλαίων στις σημαντικές ε, πιστοτικές ε, ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βελτιωθεί τον τελευταίο καιρό. Είμαστε πολύ πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσει, έχουν επίσης ανακάμψει τα κέρδη των τραπεζών, αλλά είναι σε χαμηλό επίπεδο, 4,5% ε, το 2015 και ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι δεν προβλέπονται σημαντικές βελτιώσεις για το 2016. Η αίσθηση της αγοράς, τα αισθήματα της αγοράς έχει χειροτερεύσει μέχρι τώρα το 2016. Οι τιμές των μετοχών των τραπεζών έχουν πέσει μέχρι και 30% φέτος και γενικά αποδίδουν λιγότερο από την ευρύτερη αγορά. Οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονται τόσο από την από την αντοχή των πιστοτικών ιδρυμάτων αλλά από την προοπτική κέρδους. Οι προκλήσεις στον τομέα της κυκλικής κερδοφορίας έχουν εν μέρη κατά κάποιο τρόπο μετριάσει αυτούς αρνητικούς κανόνες όπως επίσης και η σταθεροποίηση των οικονομικών συνθήκων με λιγότερες απώλειες σε επίπεδο πίστοσης. Έχουν επίσης μειωθεί και τα χρηματοδοτικά κόστη των τραπεζών μέσω της μείωσης των επιτοκίων. Έχουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε πολλές χώρες και το κόστος λειτουργίας των τραπεζών επίσης ε, υποφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις από υπερβολική ικανότητα, από υπερβολική ποσοτική μάλλον δυνατότητα. Εμείς έχουμε προχωρήσει και στο ΣΡΕΠ το 2016, μάλλον εργαζόμαστε ε, στο ΣΡΕΠ του 2016, την εποπτική δηλαδή διαδικασία και ε, αξιολογητική διαδικασία. Συγκεκριμένα αποτελέσματα πετύχαμε σαν παράδειγμα ένα υψηλότερο επίπεδο συσχετισμού ανάμεσα στα προφίλ κινδύνου και τα επιπλέον κεφάλαια τα οποία ήταν 0,26 πριν από τον Νοέμβριο του 2014 σε 0,68 το 2015. Κεφαλουχικές απαιτήσεις είναι τώρα σε παρόμοια επίπεδα και για τις σημαντικά συστημικές ε, τράπεζες της GSIB e και στους ανταγωνιστές της ε, σε άλλες δικαιοδοσίες, ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες. Εμείς χρησιμοποιούσαμε ε, μεθοδολογίες αξιολόγησης σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή επίπεδα. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν το ΣΡΕΠ το 2016. Καταρχάς εκλεπτύνουμε τη μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούμε σε σχέση με τις εσωτερικές ανάγκες κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τη ρευστότητά τους και τις χρηματοδοτικές τους δυνατότητες. Δεύτερον, βλέπουμε πώς να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε συμπληρωματικά στοιχεία όπως οι διευκρινήσεις τις οποίες έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας σε θέματα του ε, μέγιστου διανεμήσιμου ποσού όπως το λεγόμενο MDA και θέματα που σαν διευκρινιστικά έστω είναι σημαντικά για την Τραπεζική Ένωση. Είναι σημαντικό ίσως σε σχέση με το MDA να δούμε τι γίνεται και στα πλαίσια του πυλώνα 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αναλύσει το πώς θα διευκρινίσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε οι εσωτερικές λεπτομέρειες των μεγάλων εποπτικών stress test μπορούν να τροφοδοτήσουν θετικά το προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων. και επίσης το θέμα της καθοδήγησης του κεφαλαίου είναι κάτι το οποίο ε, θα είναι χρησιμαντικό και συμπληρωματικό σε σχέση με τις απαιτήσεις του πυλώνα 2. Αν ε, η καθοδήγηση σε σχέση με τον πυλώνα 2 ε, δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε, δεν θεωρείται παράληψη ή παράβαση, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω επίβλεψη και στην απέτηση επιπλέον συγκεκριμένων μέτρων έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαίων. Η καθοδήγηση του πυλώνα 2 επίσης ε, ε, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό ε, της εκκίνησης με αυτόματο τρόπο του MDA. Δεν θα χαμηλώσουμε λοιπόν τα εποπτικά επίπεδα. Οι κεφαλαιοχικές απαιτήσει είναι σε παρόμοια επίπεδα και για τις ε, τράπεζες που είναι στο εσωτερικό του SSM και για τους ανταγωνιστές τους σε άλλες ε, μεγάλες δικαιοδοσίες. Πέρα από την εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών στα πλαίσια του ΣΡΕΠ, ένα βασικό σχέδιο για την λειτουργία του SSM είναι η εναρμόνιση των κανόνων σε σχέση με τις ε, εθνικές δυνατότητες επιλογών, τα λεγόμενα OND, στα πλαίσια του CRR. Συνεχίζουμε λοιπόν την εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών και έχουμε ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για τη δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου. Η φάση αυτή φέρνει σε κατάληξη τα σχέδια για τα σημαντικά πιστοτικά ιδρύματα, προσθέτοντας ε, οκτώ περαιτέρω προβλέψεις στην ε, στον οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς πιστεύουμε ότι ο οδηγός για τα OND, για τις σημαντικές τράπεζες, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο ήδη του 2016. Για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή υψηλών εποπτικών επιπέδων και την ισότιμη λειτουργία για όλα τα πιστοτικά ιδρύματα, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές διευρύνεται η πολιτική OND και σε λιγότερο σημαντικά πιστοτικά ιδρύματα. Όταν εναρμονίζουμε όμως για μικρότερες τράπεζες, εδώ παίζει σημαντικό ρόλο ο παράγων και η αρχή της αναλογικότητας. Ε, ένα ευρύτερο τομέα, ένας ευρύτερος τομέας στον οποίο εποπτεύουμε είναι η Τραπεζική Ένωση δημιουργήθηκε η Τραπεζική Ένωση για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του πιστοτικού τομέα. Έχουν ληφθεί σημαντικά βήματα, απαιτείται όμως να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Αυτό απαιτεί πρόοδο και σε επίπεδο κατανομής κινδύνου και σε επίπεδο μείωσης κινδύνου σε σχέση με την κατανομή κινδύνου. Η ολοκλήρωση της Πιστοτικής Ένωσης απαιτεί την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος για την προστασία των καταθετών, το λεγόμενο EDIS. Το ίδις θα πρέπει να δημιουργηθεί παράλληλα με τα βήματα μείωσης του κινδύνου. Απαιτείται μια σταδιακή εφαρμογή του συνολικού μεγέθους του ίδις έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και τα εθνικά ε, συστήματα εγγυήσεων. Αυτή η σταδιακή ε, θέση σε λειτουργία θα συμπληρωθεί και από επιπλέον μέτρα τα οποία θα καταστήσουν το πιστοτικό μας σύστημα ασφαλέστερο και ανθεκτικότερο. Η μείωση των κινδύνων και η κατανομή των κινδύνων θα ενισχύσουν γενικότερα και την πιστοτική ένωση. Στον τομέα της μείωσης των κινδύνων νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ε, σε σχέση με την ε, πλήρη εφαρμογή της οδηγίας ε, για την εγγύηση των καταθέσεων και στα πλαίσια του CRR, όπως επίσης και τα MREL και επίσης το TLASC, δηλαδή τη συνολική δυνατότητα απορρόφησης ζημιών. Σε σχέση με το CRR-CRD, εδώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο, τις οποίες αναγνωρίζει η κοινοτική νομοθεσία και τις έχει χορηγήσει στα κράτη-μέλη ένας από τους τομείς τους οποίους πιστεύουμε ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι σωστές αξιολογήσεις. Το CRD4 είναι προς την κατεύθυνση αυτή μια κατελάχιστον εναρμονιστική οδηγία ε, και υπάρχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες έχουν εντοπιστεί στα διάφορα κράτη-μέλη και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, κριτήρια αξιολόγησης ε, θα πρέπει να ε, τύχουν περαιτέρω εναρμόνισης. Όταν κάποιος ε, μπορεί να αξιολογεί για διαφορετικές θέσεις σε διάφορα κράτη-μέλη, μπορεί να καταλήγει σε διαφορετικά αποτελέσματα λόγω της διαφορετικότητας και της απόκλησης μεταξύ τους των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται. Το CRR, CRD4 λοιπόν και η αναθεώρησή του θα πρέπει να εντάξουν επίσης και κάποια από τα επίπεδα τυποποίησης που έχουν προβλεφθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την ολοκλήρωση της Βασιλείας 3. Τώρα για το TILAC, για την δυνατότητα απόσβεσης ή απορρόφησης μάλλον ζημιών. Ε, νομίζω ότι το κόστος ε, της αποτυχίας ε, των τραπεζών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μοιραστεί κυρίως στους μετόχους και τους πιστωτές και όχι στους φορολογουμένους. Απαιτούνται λοιπόν ικανά επίπεδα απορρόφησης τέτοιου είδους ζημιών όταν μια τράπεζα προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτή. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του νέου MREL και πέραν τώρα της πιστοτικής ένωσης να μην ξεχνάμε τις τελευταίες εξελίξεις για τις κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη. Υπάρχει το θέμα της τιτλοποίησης, το οποίο θα συζητήσετε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια το απόγευμα. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι υπέρ των δύο νομοθετικών προτάσεων οι οποίες είναι υποσυζήτηση για τα θέματα της τιτλοποίησης τέτοιου είδους μορφές τιτλοποίησης ε, θα συνεισφέρουν σε μια καλύτερη κατανομή χρηματοδοτικών βάσεων για τις τράπεζες και θα καταστήσουν ικανή την αγορά να λειτουργήσει σωστά. Ενθαρρύνουμε λοιπόν για αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στις προσπάθειές σας. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες της ζώνης ευρώ έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητά τους, την κερδοφορία τους και την αντοχή τους. Παρ' όλα αυτά οι τράπεζες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις και σκληρές συνθήκες λειτουργίας στην αγορά. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει συγκεκριμένους <clears throat> τομείς και συνεχίζουμε την πρόοδό μας στα πλαίσια της εναρμόνισης των εποπτικών κανόνων και πρακτικών. Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του ελεγκτικού πλαισίου είναι κάτι που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ο πρόεδρος Γκουαρτιέρη, σας ευχαριστώ πολύ για την πλήρη και εκτεταμένη παρουσίαση. γρήγορα. Την εκτιμώ ιδιαίτερος. Μου άρεσε πολύ και αυτό που είπατε για τον δεύτερο πυλώνα και το MDA. Μου φαίνεται πολύ σωστή αυτή η διάκριση ανάμεσα, ανάμεσα σε guidance και requirement, σε κατευθύνσεις και σε απαιτήσεις και θα χρειαστεί ενδεχομένως, θα το δεχτείτε και σε αυτό, νομοθετική επανεξέταση και για το μέρισμα. Θα χρειαστεί να διευκρινιστεί η απόφαση αυτή. Πάντως θα υποφεληθεί η αγορά και αυτό είναι θετικό. Και για τα άλλα μεγέθη που αναφέρατε βεβαίω για το ίδιο. Τώρα, έχουμε ερωτήσει και απαντήσει. Πρώτο ο κύριος Άλβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρησή μου, καθυστέρηση πτήση μου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νούη που είναι μαζί μας εδώ. Δύο ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη αν ήδη έχετε αναφερθεί σε αυτά στην ομιλία σας. Πρώτον για την πιστοτική ένωση και τον τρίτο πυλώνα που αμφισβητείτε τόσο πολύ. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζουμε μια έκθεση για να υπάρχουν λιγότερες αμφιβολίες γύρω από τον τρίτο αυτό πυλώνα. Θα θέλαμε την όψη λοιπόν, την άποψη της κυρίας Νουή σε σχέση με τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία συνεργαζόμαστε. Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε πώς μια πιστοτική ένωση θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτό τον τρίτο πυλώνα και τι μήνυμο απαιτήσει θα υπάρξουν έτσι ώστε να μπορέσει να είναι λειτουργική η Ένωση και αυτό το κοινό ταμείο εγγύησης των καταθέσεων έτσι ώστε να υπάρχει μια αποτελεσματική πιστοτική ένωση. Να συμπληρώσω με μια ερώτηση. Δεν είναι βέβαια άμεσα αρμοδιότητά σας, σε σχέση με τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει και σε σχέση με την τιτλοποίηση. Θα ήθελα να αξιολογήσετε λιγάκι την πρόταση την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω ότι είναι θετικές οι προτάσεις αυτές. Θα ήθελα και εσείς να τις παρουσιάσετε σε επίπεδο αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΝΤΙΣ πρώτα. Ε, μας ικανοποιούν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μείωση του κινδύνου και η αναδιανομή, το resharing δηλαδή, πρέπει να προχωρήσουν ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο λόγω των διαφορετικών αφετηριών και λόγω των διαφορετικών εθνικών προγραμμάτων θα χρειαστεί να περάσει κάποιος χρόνος μέχρι να φτάσουμε σε μια ενιαία, ενιαία ε, εγγύηση ε, καταθέσεων, ευρωπαϊκή δηλαδή. Πρέπει να προχωρήσουμε ταυτόχρονα, παράλληλα, και στην μείωση του κινδύνου, risk reduction. Και οι απόπτες μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζουν τα όσα έχουν τεθεί επιτάπητος τώρα, αυτό δηλαδή το ε, αυτή τη δέσμη μέτρων για το 2020 EDIS Single Resolution Fund Backstop όλα αυτά για μείωση του κινδύνου κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό στο μεταξύ και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στόχο θα φύγουμε από την reinsurance, την αντασφάλιση, να πάμε στην co-insurance, στην συνασφάλιση μέχρι τότε για να έχουμε δηλαδή τα νότα μας καλυμμένα. Και για να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας, είμαι βεβαίω ότι ο τρίτος πυλώνας της ε, Τραπεζικής Ένωσης θα τεθεί επιτάπητος ε, μάλλον σύντομα. Οι διάφοροι πυλώνες άλλοι και αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Για την τίτλοποίηση λοιπόν, securitization, κάνουμε ε, σημαντικές προσπάθειες για να προωθήσουμε τις προτάσεις. Ε, χαιρόμαστε που προχωρεί. Ο κανονισμός θέλουμε να επιτύχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποίησης, έτσι ώστε η τιτλοποίηση να γίνει πιο ελκυστική και για τους ασφαλιστές και για τους επενδυτές, να υπάρξει από την άλλη μεριά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει ότι η διτροποίηση φέρει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που ζητούμε, δηλαδή διαφάνεια, ασφάλεια, για χαμηλά επίπεδα ζημιών ή απολειών στο διάρκεια της κρίσης. Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτόν τον τύπο τίτλοποίησης και απέναντι σε άλλους τύπους λιγότερο διαφανής τιτλοποίησης. Θα προτείνουμε κριτήρια λοιπόν για αυτή την απλή και διαφανή τιτλοποίηση, κατάλληλα κριτήρια. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνεται και συνέπειες για το τέλος που επιβάλλεται, ρυθμιστικό τέλος που επιβάλλεται στη κεφάλαια. Βέβαια, αυτό συμβαδίζει με κάποια ρωμαλαία κριτήρια που θα, ε, στη βάση των οποίων θα κρίνεται τι είναι απλή και διαφανής τίτλοποίηση και βέβαια κάτω από αυστηρή εποπτεία ε, εφόσον οι επόπτες ε, θέλουν να είναι αυστηροί και θα είναι. Υπάρχει πάντως περιθώριο για αυτή την απλή και διαφανή τίτλοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μιλήσατε για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης, δεν μιλήσατε για το τελευταίο backstop. Νομίζετε ότι πρέπει να γίνει αυτό με το έντυση ή όχι. Ερώτηση τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Brussels Economic Forum ο Klaus Regling δήλωσε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το γεγονός ότι η εποπτεία της ε, Τραπεζικής Ένωσης ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως να πρέπει να γίνει ανεξάρτητη. Διαβάζω και σε ειδήσει του Reuters ότι σκέπτονται να αφαιρέσουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εποπτικές της εξουσίες επί του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εντυπωσιακό το έργο που έχετε αναλάβει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μήπως εκεί υπάρχει κάποιο στοιχείο ανησυχητικό. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου εξηγήσετε ποια είναι η αξιολόγηση που κάνετε της δηλώσεως αυτής του ε, Προέδρου του ESM. Να μου επιτρέψετε να σας μιλήσω αγγλικά, να σας απαντήσω αγγλικά για να με καταλάβουν περισσότεροι. Σε ό,τι αφορά το backstop του ενιαίου ε, μηχανισμού του Single Resolution Mechanism δηλαδή, ε, είναι απόλυτα αναγκαίο στην δέσμη του 2020. Έχει ταχθεί λοιπόν στη δέσμη του 2020 και, και πολύ σωστά. Στο μεταξύ θα έχουμε αυτό το Loan Facility Agreement που είναι το second best για μας μέχρι να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το backstop του ενίο μηχανισμού για την ε, ρύθμιση της εξυγίανσης τραπεζών. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, εποπτεία που ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ίσως είμαι συντηρητική, εγώ πάντα έτσι το έβλεπα, ότι είναι μέρος των ε, καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως όμως να είναι καινούριο στοιχείο αυτό για τον SSM. Θα ήταν απολύτως αδύνατο να ανταποκριθούμε τόσο γρήγορα και με τέτοια ασφάλεια όπως το πράξαμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εποφελθήκαμε και εποφελούμαστε πολύ από την στήριξη που μας προσφέρουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με συστήματα ε, ηλεκτρονικής, πληροφορικής, ε, νομική στήριξη και ούτω καθεξής. Για να είμαι ειλικρινής, σε πάνω από 40 χρόνια εποπτεία που ασκώ, δεν έχω διαπιστώσει ποτέ πραγματική σύγκρουση συμφερόντων και διαρωτώ με και τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο στην περίπτωση αυτή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η νομοθεσία του SSM είναι πραγματικά ιδιαίτερα καλά φτιαγμένη από την άποψη αυτή. Βεβαίω και θέλουμε να εφαρμόσουμε και να συμμορφωθούμε απόλυτα με τον ε, κανονισμό SSM γιατί συμμετέχουν πολλές χώρες άλλωστε εκεί, αλλά είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί για να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της διακρίσεως. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο. Νομίζω θα ήταν πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε το ίδιο γρήγορα και το ίδιο αποτελεσματικά στην ανάγκη δημιουργίας του SSM αλλά τελικά, τελικά βέβαια ο νομοθέτης θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε πού θα ενταχθεί η εποπτεία. Αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπω κανένα λόγο να μην έχουμε εν τέλει την στήριξη των συναδέλφων μας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βεβαίως με διάκριση ε, καθηκόντων. Όπως ε, έχει περιλάβει και η έκθεση Μπρούγκελ, αναφέρει ε, σε αναφέρεται μάλλον σε ανεξάρτητους ε, φορείς. Το έχω πρόσφατο αυτό ε, στο μυαλό μου για το διάβαζα σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Λούκε, ευχαριστώ κυρία Νουή. Θα σας ε, μιλήσω γερμανικά εγώ με τη σειρά μου. Έχω μάλιστα πολλές ερωτήσεις και θα ήθελα να αρχίσω πρώτα με την επάνδρωση ή τη στελέχωση του SSM. Ακούσαμε περί 160 νέων θέσεων για το 2016 και έναν ακόμα ακαθόριστο αριθμό για το 2017. Αυτά όμως είναι όλα καθήκοντα που πάτε να καλύψετε, τα οποία ήταν δυνατόν να προβλέπονται από πριν. Και ε, οι επιθεωρήσεις επιτόπου και οι αξιολογήσεις εσωτερικών μοντέλων κλπ. Ποιος ελέγχει και ποιος φρενάρει εδώ την πλήρη ανάπτυξη ενός ε, οργανισμού. Οι οργανισμοί πάντοτε έχουν την τάση να αναπτύσσονται όλο και περισσότερο. Ποιος βάζει τα όρια εκεί και ποιος τραβάει το φρένο. Και ε, σημαίνει αυτό ότι θα υπάρξει αποδόμηση θέσεων στο επίπεδο των εθνικών αρχών. Βλέπω επίσης αύξηση της ε, τάξης του 25% των τελών που επιβάλλει ο SSM, που μου φαίνεται απολύτως τεράστιο. Δεύτερο, για την διαμόρφωση των αγορών κεφαλαίων και σε ό,τι αφορά την τίτλοποίηση που προωθείται, προσπαθούν να διασυνδέσουν πάλι την ευθύνη με την ενοχή. Πάλι μπαίνει εκεί όμως το θέμα του έντις και εκεί γίνεται διασύνδεση με την έννοια του risk sharing. Δεν είναι κάπως αντιφατική αυτή η εξέλιξη η τρίτη μου ερώτηση. Σας ανησυχεί ότι ενδεχομένως το έντις μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς με την έννοια ότι θα δραστηριοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους εκτός και με διαφορετικά κριτήρια από αυτές οι οποίες συμμετέχουν ήδη στην Τραπεζική Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την ε, στελέχωση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για την ε, εποπτεία είχε αποφασιστεί πριν την δημιουργία του ΙΣΣΜ και είχε αποφασιστεί χοντρικά Δηλαδή ότι ε, θα έπρεπε μετά να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Επίσης πρέπει να προσθέσω ότι διαπιστώσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πιο περίπλοκη από όσο περιμέναμε. Παράδειγμα χάρη, στο τρέχον πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας δεν υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Δηλαδή όλες οι αποφάσεις και οι πιο μικρές λαμβάνονται στο επίπεδο του Εποπτικού Συμβουλίου. Και βεβαίω ε, κάθε απόφαση συνοδεύεται από ένα σημείωμα. Γιατί αλλιώς δεν θα ξέρουν αυτοί που θα πρέπει να λάβουν την απόφαση τι θα πρέπει να κάνουν. Οπότε αυτό το γεγονός και μόνο αυξάνει πολύ το αριθμό του προσωπικού που χρειαζόμαστε για να συντάσσουν αυτά, όλη αυτή τη χαρτούρα, τα επεξηγηματικά σημειώματα. Ενώ αν λαμβάνονταν αποφάσει σε χαμηλότερο επίπεδο θα γινόταν μια απλή συζήτηση. Επίση, η έλλειψη εναρμόνιση ε, του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου είναι για μα σοβαρό ζήτημα. Παραδείγματο χάρη. Επειδή έχουμε το τμήμα εκείνο τη οδηγία το οποίο αφορά την ελάχιστη εναρμόνιση, πρέπει να έχουμε κόσμο ο οποίος θα γνωρίζει τα 19 διαφορετικά καθεστώτα και θα μπορεί να δώσει αυτές τις ε, εξουσιοδοτήσεις μέσα των 19 διαφορετικών καθεστώτων. Εάν ε, είναι πιο εναρμονισμένο το καθεστώς θα χρειαζόμαστε λιγότερο προσωπικό. Επίσης θα έλεγα ότι δουλεύουμε τόσο πολύ στη... γιατί υπάρχει εθνική διακριτική ευχέρεια. Και αυτό δεν είναι τόσο θετικό. Θα ήταν ευκολότερα τα πράγματα εάν ε, είχαμε κανονισμό που θα είχε πολύ λιγότερες και καθόλου εθνικές ε, διαφοροποιήσεις. των λεφθέντων τώρα ποιος ε, κάνει τον έλεγχο. Πρέπει να σας πω πως πρέπει να είμαστε πολύ πιστικοί ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού, της Ελεγκτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του ΔΣ της ε, Κεντρικής Τράπεζας και χρειάστηκε χρόνος βεβαίως για να μπορέσουμε να συντάξουμε αυτές τις ε, προτάσεις μας ε, γύρω στις 170 τις 170 περιπτώσεις που έχουμε εξηγήσει ήδη φέτος και γύρω στις 70 ακόμα που συντάσσονται γιατί ακριβώς ε, πρέπει στις εκθέσεις να εξηγούμε ποιες ήταν οι πιθανότητες ε, αποτελεσματικότητα σε άλλα ζητήματα. Είναι... Επίσης ένα άλλο πρόβλημα ε, μιλήσατε για τις ε, εθνικές αρχές ε, και την μείωση του προσωπικού τους. Εξαρτάται. Κάποιες είναι παρκώς τελεχωμένες, άλλες πάλι όχι. Και αρκετοί άνθρωποι οποιοι πάνε στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να ασκήσουν εποπτικό ρόλο και δεν έχουν αντικατασταθεί στις εθνικές αρχές και οι δικές μας οι αξιολογήσεις, οι απαιτήσει μας βασίζονται στο ότι οι εθνικές αρχές ε, θα έχουν τον αριθμό που μόνες τους έχουν υποσχεθεί ε, και δεν ε, το κάνουν αυτή τη στιγμή και δεν ζητάνε προφανώς αποζημίωση για πράγματα τα οποία δεν παρέχονται. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι μεγαλύτερα όργανα είναι οπωσδήποτε καλύτερα, καμιά φορά είναι λιγότερο ευέλικτα. Οπότε πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να ασκεί ο καθένας τα καθηκοντά του. Σας ευχαριστώ. Σιλβί Άκρα αριστερά, περιέργως. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση, την ταπεινή έκθεση που υιοθετήσαμε στην Ολομέλεια για τη θέση της Ευρώπης στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχουμε ανησυχίες για τον οργανισμό των ασφαλιών επίσης, όχι μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα και έχουμε και ανησυχίες για αυτά που επετοιμάζει η Επιτροπή της Βασιλείας. Αυτό που λέγει η έκθεση και δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη, προφανώς και απαιτείται να υπάρχει πλήρης ισοτιμία και δικαιοσύνη σε επίπεδο ανταγωνισμού. Προφανώς και πρέπει να υπάρξει ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, αλλά από πού παίρνει την νομιμότητα που απαιτείται η Επιτροπή της Βασιλείας, έτσι ώστε να προσθέσει τόσα στοιχεία στα συμπεράσματα και βέβαια τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν ότι έγιναν σημαντικά βήματα προόδου, αλλά από εδώ και πέρα πώς βλέπετε εσείς αυτό το κύμα το μεγάλο το οποίο θα μας στείλει η Επιτροπή της Βασιλείας. Πώς μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε σε μια εποχή χαμηλής ανάπτυξης, όπου η απασχόληση είναι ανεπαρκέστατη, να σφίξουμε ακόμα περισσότερο στις ροές κεφαλαίων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ευνοηθούν επιστοτικοί ε, τομείς άλλων περιοχών του κόσμου και δεν θα προσδώσει περαιτέρω σταθερότητα στο δικό μας. Θα συνεχίσω στην Αγγλική, λέει ακάθεκτη η κυρία Νουή. Εμείς πράγματι έχουμε μία εντολή, έχουμε όρους αναφοράς που έχουμε δώσει συγκεκριμένα στην Επιτροπή της Βασιλείας. και εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το SSM, με τμήμα εμπασπεριτώσει αυτής της ομάδας και εγώ, όπως επίσης και ο Βίκτορ Κωνστάνσιο και συμμετέχει πολλές φορές και ο κύριος Ντράγκη, ο πρόεδρος. Η Ευρώπη εκπροσωπείται εμπασπεριτώσει με καλό τρόπο και η εντολή είναι επίσης σαφής. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις κεφαλαιοχικών απαιτήσεων στον τομέα του πυλώνα 1 ίσως κάποιες διευκρινήσεις να οδηγήσουν στην αύξηση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Αλλά συνολικά τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των κεφαλαίων. Ταυτόχρονα αναγνωρίζω ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αντιμετωπίζονται τίνουν κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται να τίνουν προς μία και μόνη κατεύθυνση. Αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλής και από την νέα τυποποιημένη αντιμετώπιση η οποία θα πρέπει να είναι ευαίσθητη σε κινδύνους και πώς μπορούν οι ροές και ε, οι, ε, τα επίπεδα προστασίας να υπολογιστούν με σωστότερο τρόπο. Πάντως έχει υπάρξει μια ε, τεράστια πλειοψηφία έτσι ώστε να μην υπάρξει σημαντική αύξηση των απαιτούμενων κεφαλαίων και δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτό και δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Είδα κάποιες προτάσεις ε, έρευνας από ορισμένα πιστοτικά ιδρύματα που αναζητούν μια διαφορετική ρητορική. Όμως ταυτόχρονα θα μπορούσα να πω ότι στην ουσία αναλύουν με πολύ ε, συγκεκριμένο τρόπο τις δυνατότητες ε, εξελίξης. και αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σημαντική αύξηση, αλλά είναι μια πολύ επιμέρους λογική η οποία δεν είναι στο εσωτερικό της εντολής που έχει δοθεί στην Επιτροπή της Βασιλείας. Προσωπικά εγώ έχω κι άλλο ένα λόγο για να είμαι σαφής στον τομέα αυτό. Εγώ θέλω χώρο για τις κρίσεις των αυτών οι οποίοι επιβλέπουν Θέλω περισσότερο χώρο στα πλαίσια του πυλώνα 2. Συνεπώς λοιπόν εμείς ε, είμαστε διατεθειμένοι ε, να προχωρήσουμε στα πλαίσια της εποπτικής πρότασης την οποία κάνει η λεγόμενη Ghost Group. ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι ως ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα ε, και με εσά και ίσως και με την Επιτροπή της ε, Βασιλείας. Αμέσως. Λοιπόν, Φάμπιο Ντεμάζη. Σας ευχαριστώ. Κύριε για τα όσα είπε η κυρία Μπερές για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της εποπτείας των τραπεζών και της νομισματικής πολιτικής. Εγώ καταλήγω σε διαφορετική αξιολόγηση. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση του Unintelligence και τα έγγραφα που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία δεν μπορούμε να σχολιάσουμε βεβαίως, ε, είναι κάπως ε, διαφορετική η δικιά μου εξελόγηση. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω πως εσεί εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την Hansa Nordbank από την πόλη μου, το Αμβούργο. Η Κομισιόν αποφάσισε πως η Hansa Nordbank ε, μπορεί να εγγράψει στα βιβλία της ε, το πολύ 6,2 ευρώ για να αγοραστούν από τα, κρατηδια, τα κρατήδια του Αμβούργου και του Σλέσφι Χόλσταϊν. Και αρχές ε, Μαρτίου μετά, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, η Κομισιόν μίλησε για ε, μια έκπτωση 60% αυτό όμως σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ του Αμβούργου σημαίνει πως ε, οι έλεγκτες της τράπεζας είπαν πως κινδυνεύει πλέον η ίδια η ύπαρξή της. Και υπάρχει άρα κίνδυνος και υπήρξε μία έγκαιρη περιοδοποίηση για το ίδιο κεφάλαιο της ε, τράπεζας, καθώς υπάρχουν μόνο 5 δισεκατομμύρια τα οποία μπορούν να εγγραφούν με ένα ποσοστό του 50%. Θεωρείτε λοιπόν πως με αυτό το παζάρι υπάρχει κίνδυνος για την ανεξαρτησία των τραπεζών. Δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω τι άποψη έχετε για αυτά τα οποία αναφέρουν τα ΜΜΕ για την Γαλλία και την Ιταλία όπου οι απαιτήσει ιδίων ε, κεφαλαίων θα πρέπει να είναι πάνω από το 8% εκτός από περιπτώσεις ανάγκης και επίσης ε, το τίλακ θα μπορέσει να μετατραπεί σε μετοχές. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει μια χαλάρωση των κανόνων τους οποίους είχαμε αποφασίσει. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αναφέρατε ότι εγώ δεν θα αναγνωρίσω δημοσίως ε, κάποια σύγκρουση συμφερόντων, ε, ούτε ιδιωτικό. Ε, δεν έχω συναντήσει τέτοια περίπτωση. Βεβαίω, ίσω είμαι προκατηλημένη. Αυτό το αναγνωρίζω, γιατί πρόκειται για ένα καθεστώ το οποίο είναι νέο, αλλά ειλικρινά νομίζω πως τα πάντα έχουν γίνει στον σχετικό κανονισμό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Και εντάξει, Γνωρίζω πως ελέγχομαι αυστηρά και δικαίως. Η Αντιπρόεδρος, η Γερμανίδα συνάδελφος ε, έχει ανατραφεί σε διαφορετικό περιβάλλον ε, και νομίζω πως έχουμε βρει μια καλή ισορροπία. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας δεν μπορώ να σχολιάσω για μεμονωμένες συγκεκριμένες τράπεζες. Τούτου λεχθέντος, οι εποπτικές αρχές δεν ε, καθορίζουν ε, ε, τα νούμερα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμείς παρέχουμε συνέπεια, ίσους όρους ανταγωνισμού. Βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξετάμενο πλαίσιο. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν τράπεζες ε, οι οποίες ε, είχαν συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσει. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες άρα, που πάνε με το σε αυτό και συμμορφωνόμαστε. Φροντίζουμε και οι τράπεζες να συμμορφώνονται. Έτσι, θα, έτσι ήταν και πριν από το μηχανισμό των εποπτικών και μετά. Ναι, για το TILAC. Ε, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι εν εξελίξη. Ειδικά μεταξύ έμρελ και TILAC και το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη έτσι ώστε οι τράπεζες να μην έχουν περισσότερους περιορισμούς από τους ανταγωνιστές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαι σίγουροι πως ε, είναι κάτι το οποίο θα δει το Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο κάτι στο οποίο πρέπει να απαντήσει η συνάδελφος η Ελκε Κένιγκ για την σχέση μεταξύ Έμρελ και Τίλακ. Για να προχωρήσει ακριβώς ε, η υπόθεση του Έμπρελ. Σας ευχαριστώ. Και οπωσδήποτε θα το κάνουμε αυτό λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε δηλαδή ως Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Φίλιπ Λάμπερτς. Τέσσερις γρήγορες ερωτήσεις και μπορείτε να απαντήσετε τηλεγραφικά. Πρώτον, λέγεται ότι η μη ικανοποίηση σε σχέση με τον πυλώνα 2 Φαίνεται ότι οι απαιτήσει του πυλώνα 2 δεν είναι λιγότερο δεσμευτικές από ότι του πυλώνα 1, οπότε η ερμηνεία η οποία, η οποία δίδεται μου είναι ακατανόητη. Συμφωνείτε με την κυρία Κέρνινγκ που λέει ότι θα πρέπει ε, να βάλουμε ένα ποσοστό του MREL γύρω στο 8%. Τώρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παιδευόμαστε με αυτό εδώ και 10 χρόνια. Μήπως θα πρέπει, εν πάση να σπάσουμε το απόστημα. Να βρούμε έναν τρόπο, εν να σταματήσει η ανασφάλεια σε σχέση με τον τομέα αυτό. Και τέλος, για τον μηδενικό κίνδυνο σε σχέση ε, με τον κίνδυνο που προκαλείται από το δημόσιο χρέος ε, αυτό μπορεί να συνεχίσουμε να το κάνουμε εφόσον κάθε πιστοτικό ίδρυμα έχει ένα χαρτοφυλάκιο σταθμισμένο τίτλων του δημοσίου. Αν μια τράπεζα, σαν παράδειγμα, έχει τέτοιες, τέτοιους τίτλους μοιρασμένους και σταθμισμένους σωστά, τότε μόνο να είναι μηδενικός ο κίνδυνος. Τηλεγραφικά λοιπόν πάντα σχετικά με τον πυλώνα 2. Οι διευκρινήσεις τις οποίες έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ζητήσαμε να υπάρξει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν διαφορετικά συστήματα για να καθοριστούν οι απαιτήσει του πυλώνα 2 σε σχέση με τους εμπλεκομένους και του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2 και ε, τους, ε, τις γραμμές προστασίας. Έχουμε τη συμμόρφωση με το MDA αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κέρδος εφόσον δεν υπάρξει σεβασμός και επίσης η καθοδήγηση του πυλώνα 2, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με το MDA. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, εμείς περιμένουμε από τα πιστοτικά ιδρύματα να λάβουν υπόψη αυτά που είπα και να μην παραβιάσουν την καθοδήγηση την εποπτική. Είναι κάτι το οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ένας καλός τρόπος έτσι ώστε να διατηρήσουμε το επίπεδο του κεφαλαίου. Απαιτείται κάποιος χρόνος έτσι ώστε η καθοδήγηση να γίνει πλήρης απέτηση, η οποία ε, επηρεάζεται εν πολλής από τις ε, συνθήκες και προϋποθέσεις ε, του CRD4. Πάντως το υλικά πιστεύουμε ότι θα απαιτηθεί να διατηρηθεί το επιθυμητό επίπεδο κεφαλαίου στο σύστημα σχετικά με το MRL. E Τι είναι αυτό το 8% που είπατε. Αν θεωρήσουμε δεδομένη τη σύγκριση ανάμεσα στο MRL e και το TILAC, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε από τη μία το 6% συν. Με ό,τι ακολουθεί μετά το 6% έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα σύγκρισης. και έτσι να μπορούμε να εφαρμόσουμε το τύλακ για τα ευρωπαϊκά πιστοτικά ιδρύματα. Προφανώς δεν μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα από τις μεσαίες και μικρές ε, τράπεζες από ό,τι ζητάμε από τις ε, σφαιρικές μεγάλες, ε, μεγάλου βάρους. Ταυτόχρονα το 8% αυτό συνδέεται πάρα πολύ συχνά με τις ε, ζημίες και τα bail-in που μπορεί να προβλέπονται από το Ταμείο για την Επίλυση των Τραπεζών. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι την εγγύηση των εγγύησεων. Οτιδήποτε υπάρχει λοιπόν μέχρι τις 100.000 είναι θεωρητικά χρησιμοποιήσιμο για τα Μπέιλιν. Από την άλλη για τα Τίλαξ θα δούμε τι θα πει ο νομοθέτης όταν μιλάμε ε, για τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, τότε τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά εδώ. Στόχος πάντως είναι το 8% είτε του MREL είτε του μπειλιν, είναι η ανακεφαλαίωση των σωστών τραπεζών, των ορθών τραπεζών, μετά από την παρέμβαση. Ελπίζοντας και διευκρινίζοντας ότι έχουμε να κάνουμε με μια καλή τράπεζα, δηλαδή καλύτερη από την προηγούμενη, οπότε θα έχει μικρότερες κεφαλουργικές ανάγκες. Διότι το κακό κομμάτι θα έχει πλέον εξαιρεθεί, αφαιρεθεί. Τώρα για το δημόσιο χρέος το 0 βαθμός κινδύνου. Νομίζω ότι οι νομοθέτες θα είναι αρκετά σοφοί έτσι ώστε να βρούνε τη σωστή λύση. Ίσως να είναι και τμήμα του πακέτου 2020. Εγώ βλέπω κάποιες προτάσεις οι οποίες συνδυάζουν την ποιότητα του δημοσίου χρέους από τη μία και τη συγκέντρωση από την άλλη. Είναι ευφυής αυτή η λογική. Θα δούμε τι θα γίνει. Σε σχέση τώρα με τις μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις, δάνεια. Και εδώ βρισκόμαστε σε φάση επεξεργασίας και μέσω μιας συμπληρωματικής επιστολής θα σας μεταφέρουμε τις απόψεις μας έτσι ώστε να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Αυτό το 8% θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας, λέει ο κ. Γουαλχέρη. Το 44 είναι διαφορετικό από το 45 έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε. FDD δεν θέλει κάποιος το λόγο. Α, όχι, ο κύριος Μονό και το INF. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Νουή, δύο ερωτήσεις. Αν ανασυνθέσουμε το Ευρωπαϊκό Οργανικό Πάνελ βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια σχιζοφρένεια. Από τη μία το ESM και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SSM συγγνώμη, και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία το SSM ασχολείται με τη χαμηλή αποδοτικότητα των τραπεζών, από την άλλη η τράπεζα με τα χαμηλά επιτόκια χαμηλώνει ακόμα περισσότερα τα κέρδη των τραπεζών και εμεί επιτρέπουμε να λειτουργούν όλες αυτές ε, οι εταιρείε αξιολόγηση με αμφισβητούμενα συστήματα και τα χρησιμοποιείτε και εσείς σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι δεν θα λύσετε τα προβλήματα βέβαια των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ταυτόχρονα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μπλοκάρει τις πιο ευφυείς αντιμετωπίσεις ε, για να καταπολεμήσει το δημόσιο χρέος. Η Ιταλική κυβέρνηση έχασε ένα χρόνο λόγω των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι καταθέτες λοιπόν και οι επενδυτές είναι ανήσυχοι σε σχέση με τις ομολογίες και τις καταθέσεις που έχουν. Τα πράγματα λοιπόν, ιδιαίτερα σε σχέση με τους λεγόμενους κοινού τίτλους, όπως επίσης και το MREL. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα επηρεάσει όλα αυτά θετικά. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι εθνικές αρχές που ασχολούνται με θέματα πρόληψης, δεν νομίζω τώρα για τις ελληνικές τράπεζες. Ενώ η κεντρική τράπεζα ελέγχει πλέον και είναι κηδεμόνας, βλέπουμε να υπάρχουν πάντα και μετά από το νέο πρόγραμμα χρηματικής βοήθειας προς την Ελλάδα προβλήματα στις τράπεζες αυτές αν δεν μπορέσατε να μειώσετε τις αμφισβητούμενες, μη εξυπηρετούμενες ε, δανειακές υποχρεώσεις, ε, τότε τι θα κάνετε για τις υπόλοιπες τράπεζες στην Ευρώπη. Euh, ε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν βλέπω κάποια συμβατότητα στον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Νομίζω ότι σε πλήρη συμβατότητα με τις αρχές ε, του διαχωρισμού, εμείς ε, σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθούμε τα πράγματα για να βοηθήσουμε την οικονομική κατάσταση και όσο μας αφορά εμείς κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, να είμαστε καλοί επόπτες σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τα πιστοτικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα το κόστος της χρηματοδότησης των τραπεζών έχει μειωθεί μέσω των πολιτικών μας. Η πιστοτική ποιότητα των ισολογισμών και των απολογισμών έχει και αυτή βελτιωθεί και οι δανειστές είναι σε καλύτερη θέση για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα δάνεια, τα χρήματα μάλλον. Οι τράπεζες είναι δυναμικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν ε, αντίξωες συνθήκες σε δύσκολα περιβάλλοντα, χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλός πληθωρισμός είναι κάτι που καθιστά τα πράγματα πιο περίπλοκα, πιο δύσκολα για την οικονομία, αλλά όχι μόνο και για τα πιστοτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, για τις τράπεζες να αξιολογήσουν την βιωσιμότητα του μοντέλου του επιχειρηματικού τους και να καταστούν πιο αποδοτικές. Υπάρχουν περισσότερες ε, ε, δυνατότητες για τις τράπεζες αυτές, το κόστος λειτουργίας τους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουν, πώς μπορεί να βοηθηθεί και να γίνει χαμηλότερο. Η ψηφιοποίηση επίσης είναι κάτι το οποίο να μην χρησιμοποιείται μόνο για όλους τους πελάτες. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι θέλουν και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω ψηφιακά μέσα, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία που θα μπορούσαμε. Πάντως, η αβεβαιότητα την οποία, ε, στην οποία αναφερθήκατε είναι ο χρόνος που απαιτείται για να υπάρξει μια σωστή νομοθετική επεξεργασία και πρόταση. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό έχουν προχωρήσει με τρομακτική ταχύτητα. Ο κανονισμός του SSM, σαν παράδειγμα, ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Είναι κάτι το πάρα πολύ σύντομο. Σχετικά τώρα με τις μη εξυπηρετούμενες ε, εκθέσεις, δάνεια. Και αναφερθήκατε και στις ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες κάνουν αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από πλευρά των οργάνων. Και προς το παρόν δεν έχουν καθυστερήσει. Το Hellenic Stability Fund, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώ επίτηδες ε, αυτό τον όρο, κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει με τους επόπτες της Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, για να προχωρήσουν επίσης και στην αντικατάσταση με τους καταλληλότερους και τα πιο ε, καλά στελέχη των διοικητικών του συμβουλίων. Λοιπόν, συμβουλίων. Ε, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό. Ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει και γίνεται. Thank you, José Manuel Fernández. Obrigado, Presidente. Madame σε ευχαριστώ, José Manuel Fernández. Σε ευχαριστώ, κύριε Νίγη. Κοιτάξτε, έχετε την Προεδρία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και άρα εποπτεύετε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και άρα την και ε, General de Depositos, τη μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας. Τώρα, η κυβέρνηση θα δώσει λεφτά των φορολογουμένων στην ε, τράπεζα αυτή ε, μιλάμε για ποσά των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποια είναι λοιπόν η θέση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για αυτή την ε, κατάσταση και την κίνηση. Ε, τέσσερα, με συγχωρείτε. Τέσσερα Πώς φτάσαμε σε αυτή την ε, κατάσταση και σε αυτά τα ποσά. Κοιτάξτε. Ε, το μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο είναι πάντα θετικό για την εποπτική αρχή και για την κατάσταση των τραπεζών. Τώρα δεν θα αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αν μια τράπεζα είναι δημόσια τράπεζα και αυτός ο οποίος έχει το μετοχικό κεφάλαιο είναι το κράτος, προφανώς όταν η τράπεζα χρειάζεται στήριξη μέσω μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να παρεμβεί το κράτος σε αυτή τη φυσιολογική κατάσταση για μια μεγάλη τράπεζα. Τούτου λεχθέντος η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξετάζει προσεκτικά τέτοιε ε, περιπτώσεις. Οι δημόσιε τράπεζες δηλαδή που απαιτούν περαιτέρω ρευστότητα από το κράτος ε, πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι κερδοφόρες και ότι πρόκειται για φυσιολογική επένδυση ενός ε, μετόχου στην τράπεζα και όχι κρατική ενίσχυση. Ε, δεν θέλω τώρα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτός κανόνας ισχύει για την Πορτογαλία, για τις δημόσιες τράπεζες στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες. Το ίδιο ισχύει. Εάν μια δημόσια τράπεζα χρειάζεται επιπρόσθετα κεφάλαια, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν θα φροντίσει να διαπιστώσει ότι είναι κανονικές επενδύσεις και όχι κρατικές ενισχύσεις. Αυτά δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω. Σας ευχαριστώ κυρία Καϊλή. Thank you. Thank you, sir. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Νουή. Όλοι ξέρουν πως ε, τα κίνητρα των ε, τραπεζών για να βγάλουν κέρδη υπερβαίνουν το κίνητρο για υπεύθυνη συμπεριφορά. Ε, βλέπαμε το τι έγινε και σε διάφορες χώρες όπου είχαν μια κουλτούρα της αγοράς και ασθενείς ε, θέσμους. Οι εσωτερικές δομές ε, διακυβέρνησης των τραπεζών και η ικανότητα των εποπτικών αρχών για έλεγχο της αγοράς επέτρεψαν στους τραπεζίτες, όπως ανεφέρατε ήδη, και σε άλλους ενδιάμεσους να θεωρούν ότι ε, μπορούν να αυξήσουν τα, τα κέρδη τους ε, μέσω υπερβολικών κινδύνων, υπερέκθεση σε ρευστότητα και προβλήματα φερεγγιότητας και τελικά καταλήξαμε στην παγκόσμια οικονομική κρίση και την κρίση της Ευρωζώνης. Και βεβαίως ο κίνδυνος ε, είναι κίνδυνος και ενίσχυσης της οικονομικής συγκυρίας ε, και υπάρχει και κινδύνος μετάδοσης και δεν έχει ακόμα ο μηχανισμός σας αντιμετωπίσει το θέμα της ε, διαφορετικής ποιότητας της εποπτείας των τραπεζών σε όλα τα 28 κράτη-μέλη και τη διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου. Πρόκειται για ένα στοιχείο κρίσιμο γιατί η επιτυχία του μηχανισμού σας ε, εξαρτάται από την διαχείριση αυτών των διαφορών όπως αναφέρατε. Και στην περίπτωση της Ελλάδας οι διαδικασίες εξέταση των εποπτικών μηχανισμών και καταλληλότητας των τραπεζών ήταν ανεπαρκείς καθώς είχαμε γεγονότα τα οποία ε, γεγονότα ανάληψη κινδύνου τα οποία ακόμα δεν έχουν επαρκώς ε, ερευνηθεί. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής πώς σκοπεύει ο μηχανισμός σας να δει ζητήματα έπρεπους ε, συμπεριφοράς ε, δεδομένου του ότι έχει μεγάλη σημασία ο τραπεζικός κλάδος για την ε, ανάπτυξη και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε τους πολίτες οι οποίοι πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν τις επανειλημμένες ανακεφαλαιοποιήσεις. Και η δεύτερη μου ερώτηση. Σκοπεύετε και αν ναι πώς να περιλάβετε στα stress ε, test μηχανισμούς αξιολόγησης ε, του επιχειρησιακού κινδύνου που δύσκολα ποσοτικοποιείται. Κοιτάξτε, κίνδυνος τώρα απρεπούς συμπεριφοράς ή Ε, επιχειρησιακή κίνδυνη. τα ε, αυτά είναι πέρα από τον ευρωτικό ρόλο, φορούν προφανώς τους νόμους στην κάθε χώρα, αλλά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που διατρέχουν στις ε, περιπτώσεις αυτές και το λαμβάνουν αυτό υπόψη στον ορισμό του κεφαλαίου κινδύνου και βεβαίως ε, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός. Του τελευταίντος, βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από σωστούς ε, εσωτερικούς ελέγχους ε, και Βεβαίω και εμείς θα πρέπει να προχωράμε την έρευνα εις βάθος όταν ε, έχουμε τράπεζες οι οποίες ε, θεωρούμε ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες. Στο παρελθόν αυτό αφορούσε λειτουργίες ε, στην αγορά, αλλά τώρα πλέον με το περιβάλλον αυτό του Μπέιλιν θεωρώ πως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος παντού. Δηλαδή θα πρέπει οι τράπεζες να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους οποίους πουλάνε, οι επενδυτές που αναλαμβάνουν κάποιες ε, εκθέσεις ε, να είναι ενήμεροι για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Αναφέρατε τις ελληνικές τράπεζες. Δεν βλέπω ο αυτός να είναι ο σημαντικότερος για τις ελληνικές τράπεζες. Ε, προφανώς υπάρχει κίνδυνος, αλλά όχι αυτός. Δεν νομίζω να είναι αυτός ο σημαντικότερος. Λοιπόν, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ, Brian Hayes. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ανοή, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα του κινδύνου που φίξατε στην παρουσίασή σας, το ότι πρέπει να αντιληφθούμε πού βρίσκεται αυτός ε, εντός ε, του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος ειδικότερα. Αλλά δεν θα σας ζητήσω να σχολιάσετε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα που έχουν σημαντική έκθεση στην Βρετανική αγορά, δηλαδή το Brexit. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μάθω τι έχει κάνει το SSM μέχρι στιγμής για να τονίσει αυτόν τον κίνδυνο σε τράπεζες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη Βρετανική αγορά και στην χώρα μου, την Ιρλανδία και αλλού. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο μηχανισμό έχουν έρθει σε επαφή με τράπεζε στην Ιρλανδία και αλλού για να μάθουν κατά πόσο είναι έτοιμε για πιθανό Brexit δεδομένη της έκθεσης που υπάρχει για καταθέτες, επενδυτές κτλ. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια αξιολόγηση για το πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες ε, στους τομείς όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Και δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε υπάρχουν σχέδια ανάγκης για να αντιμετωπιστεί αυτή η πιθανότητα. Με την έννοια ότι θα είμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό εποπτικό περιβάλλον σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε. Και τέλος, θεωρείται ε, προτιμότερο οι τράπεζες ε, να κάνουν αυτό το οποίο έκανε η JP Morgan και άλλοι, δηλαδή να δημοσιεύουν ε, την άποψή τους για το τι σημαίνει ένα πιθανό Brexit. Δηλαδή έχει δικαίωμα ο κόσμος να γνωρίζει το τι έχουν κάνει οι τράπεζες ως σχεδιασμό ανάγκης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολη ερώτηση βέβαια σχετικά με την Βρετανική έξοδο. Δεν θα προσπαθήσω βέβαια να προβλέψω τίποτε ούτε καν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ε, εξόδου της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα, για την εποπτεία. Εμείς είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού που προετοιμάζεται, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για αυτό το ενδεχόμενο. Για αυτή την ενδεχόμενη έκβαση του δημοψηφίσματος. Και σε ό,τι αφορά την εποπτική λειτουργία, αυτό γίνεται βεβαίως ανά τράπεζα. Για κάθε τράπεζα που είναι πιθανό να υποστεί συνέπειες, προβαίνουμε σε ανάλυση από το GST, το Joint Supervisory Team, σχετικά δηλαδή με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, ζητούμε τα σχέδια των τραπεζών που βέβαια είναι διαφορετικά μεταξύ τους ανάλογα με τον ενδεχόμενο κίνδυνο και με την ενδεχόμενη επίπτωση που θα πρέπει να καλυφθεί. Και βέβαια αξιολογούμε τα σχέδια αυτά, τα βάζουμε σε δοκιμασία σχετικά δηλαδή με το τι επιπτώσει θα έχει η εφαρμογή του στην αγορά. Αυτό είναι λίγο πολύ business as usual. Οι τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες για την αντιμετώπιση ενδεχομένων. Είναι σωστό να γίνει και ένα τέτοιο εγχείρημα πριν από ένα ενδεχόμενο Brexit, ώστε να είμαστε ικανοί και ικανές ε, για να αντιμετωπίσουμε την αναταραχή που μπορεί να προκύψει. Αυτό είναι και καλή εκπαίδευση για τις τράπεζες και με την έννοια αυτή είναι καλοδεχόμενη η άσκηση αυτή. Θα δούμε ποια θα είναι τελικά η έκβαση και θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσουμε τις... αυτά που κάνουμε δηλαδή και να τα εφαρμόσουμε και σε άλλους. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Πέτερ Σίμων. Κυρία Νουή, αξιότιμη κυρία Νουή, βρίσκομαι εδώ δύο ερωτήσεις. Και οι δύο για πράγματα που ε, αναπτύξατε προηγουμένως. Έχω μία πρώτα βασική, ας πούμε, ερώτηση αρχής. Είπατε για το έντις κατανομή του κινδύνου και μείωση του κινδύνου. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ποια μέτρα μείωση του κινδύνου θεωρείται αναγκαία για την ύπαρξη του έντις. Δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην διαμόρφωση της εποπτείας που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξηγήσατε εσείς προηγουμένως γιατί έγινε αυτό, γιατί υπήρχε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι που παρακολουθήσαμε τα πράγματα είδαμε πόσο ταχύτατη ήταν η ανάγκη να αντιδράσουμε, πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη να αντιδράσουμε ταχύτατα τότε. Τώρα, ο Ιγνάτιο Αντζελόνι στην Φραγκφούρτη σε μια τοποθέτηση που έκανε τον Μάρτιο δήλωσε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν συμβατικές βάσεις για μια ανεξάρτητη εποπτεία, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε τέτοιους προβληματισμούς και πώς βλέπετε την προοπτική για ε, την εγκατάσταση αυτής της αρχής. Υπάρχει απόφαση να τοποθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί. Εάν ναι, μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Κύριε Νουή, σε ό,τι αφορά risk sharing και risk reduction, γνωρίζω ότι το κόψιμο του ομφάλιου λόρου μεταξύ του δημόσιου χρέους και και των τραπεζών είναι στα χέρια του νομοθέτη. Και σωστό είναι αυτό. Καλωσορίζω λοιπόν τα μέτρα που θα ληφθούν στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θα έλεγα γενικά να γίνουν πιο υγιείς και πιο ασφαλείς οι τράπεζες. Αυτό είναι το βασικό καθήκον μου. Αν κάνω δηλαδή τη δουλειά μου σωστά, η μείωση του κινδύνου θα επέλθει και μόνο με την ορθή εποπτεία και νομίζω ότι ήδη συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά το ενδεχόμενο στο μέλλον, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή των συνθήκων, μπορεί να έχουμε ανεξάρτητη τραπεζική εποπτεία, ίσως. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να προκαλέσουμε την αλλαγή αυτή. Εγώ πιστεύω όχι. Εγώ νομίζω ότι καλά είμαστε όπως είμαστε τώρα. Όμως ο νομοθέτης είναι εκείνος που θα αποφασίσει. Για την ώρα είναι τόσο επιτυχής η έκβαση της προσπάθειάς μας να παραμείνουν οι τράπεζες ασφαλείς, ώστε κανείς δεν αλλάζει κάτι που λειτουργεί, που αποδίδει. Εάν δεν είναι επαρκής η επιτυχία, τότε μπορεί να υπάρξει η αλλαγή αλλά νομίζω ότι καλά τα πάμε και η προσπάθειά μας αυτή είναι. Αλλά, ξαναλέω, ο νομοθέτης αποφασίζει και ίσως θελήσει να τοποθετήσει την εποπτεία σε άλλο πλαίσιο. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η ποιότητα της εποπτείας. Να επανέλθω. Για το έντις κατάλαβα καλά ότι είπατε ότι για τα μέτρα μείωσης του κινδύνου, αυτά που έχουν δρομολογηθεί δηλαδή, δεν χρειάζονται άλλα και ότι τα υποστηρικτικά μέτρα που λαμβάνονται αρκούν ή χρειάζονται και άλλα πρόσθετα μέτρα μείωσης του κινδύνου. Δεν είπα αυτό. Risk reduction είναι μουσική στα αυτιά των εποπτών. Οποιαδήποτε μείωση κινδύνου για μας είναι καλό πράγμα. Είμαι βεβαία ότι ο νομοθέτης θα λάβει και άλλα μέτρα. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τον τρίτο πυλώνα της ε, Τραπεζικής Ενώσεως. Χρειαζόμαστε τον νέο μηχανισμό για τα ε, προγράμματα ε, εγγύησης καταθέσεων θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή μείωση του κινδύνου κάνοντας πιο υγιείς και πιο ασφαλείς τις τράπεζες. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα μείωσης κινδύνου και είμαι βεβαία ότι ο νομοθέτης θα αποφασίσει και εμείς βεβαίως θα πράξουμε ανάλογα με τις αποφάσεις του. Ευχαριστώ και εμείς εδώ, δηλαδή ο παρόν νομοθέτης έχει ήδη εκφράσει άποψη. Υπάρχει θέση μας λοιπόν γι' αυτό. Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδης και πάλι. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι Έχουμε ήδη καταθέσει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά άλλα 4. Έχουμε δεσμεύσει δηλαδή τα κεφάλαια αυτά. Διαρωτώ με. Δεν σημαίνουν αυτά αποτυχία του εποπτικού μηχανισμού. Είναι φυσικό να χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι με τέτοια ποσά και κανείς τελικώς να μην αναλαμβάνει ευθύνη. Ευχαριστώ. Έχω κι άλλη μια ερώτηση. Εσείς είχατε ανάμειξη στην εξυγίανση, τραπεζική εξυγίανση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2015. Σας άσκησαν κάποια στιγμή οι κυβερνητικές αρχές της Πορτογαλίας πίεση για να βρείτε λύση στο πρόβλημα της ε, τράπεζας Μπάνιφ στην ε, Πορτογαλία πριν από το τέλος του 2015 για να μην μεταφερθεί το πρόβλημα το 2016 σας άσκησαν πίεση οι πορτογαλικές αρχές. Είχατε προηγούμενες επαφές με την Σανταντέρ ή με άλλες τράπεζες σε σχέση με την τράπεζα Μπάνεφ. Ήρθατε εσείς σε επαφή με τις πορτογαλικές αρχές ή όχι για να τους ζητήσετε να εξετάσουν και άλλες δυνατότητες ή εργαστήκατε μονάχα με την Σανταντέρ και υπήρχε νομική βάση ώστε να αναμειχθεί η τράπεζα Σανταντέρ με τον τρόπο που ανεμίχθη. Για το πρώτο θέμα που είπατε δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά την Πανίφ είναι απλό. Δεν επόπτευσα εγώ την τράπεζα αυτή, δεν την γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τα μέτρα που έλαβε η Εποπτική Αρχή για, την σχετική, τη συγκεκριμένη τράπεζα. Η μόνη δράση που ανέλαβα σχετικά ήταν μία ημέρα στη διάρκεια της αδείας μου έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Υπουργό Οικονομικών της Πορτογαλικής Κυβέρνησης που μου είπε δεν καταλαβαίνω τι μου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι εννοούν. Αυτό προσπάθησα εγώ να το εξηγήσω. Τι θεωρούσα ότι εννοούν γιατί έχω ε, πιο συχνά επαφές βέβαια με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής από ότι ο Υπουργό Οικονομικών. Του είπα όμως για να είμαι και σίγουρη θα τηλεφωνήσω στην Κομισιόν. Τηλεφώνησα στην Κομισιόν και μου επιβεβαίωσαν ότι οι εξηγήσει που έδωσα στον Υπουργό ήταν ορθέ. Ε, επιβεβαίωσα λοιπόν στον Υπουργό αυτά τα πράγματα. Μετά από την επιβεβαίωσή μου, ο Υπουργό μου είπε εάν πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζω κάτι άλλο, διότι εγώ του είπα ότι η Κομισιόν θα μου πει, εμένα δηλαδή, εάν υπάρξουν νέες εξελίξεις. Και να μου πείτε όσο, όταν ενημερωνόμουν λοιπόν από την Κομισιόν για τις νέες εξελίξεις, έστελνα και ένα email στον Υπουργό για να του εξηγώ πράγματα που θεώρησα ότι θα τον ενδιαφέρουν. Και αυτά τα email δημοσιεύτηκαν. Μπορεί να τα δει κανεί δηλαδή, είναι δημοσιοποιημένα. Δεν έχω απολύτως καμία επαφή με την Santander, και ούτε δέχθηκα πίεση από οποιονδήποτε για να κάνω οτιδήποτε. Ξαναλέω, δεν επόπτευα τη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν συμμετέσχουν στην συγκεκριμένη εξυγίανση, απλώς μετέφερα μια εξήγηση που μου ζήτησαν. Και όλα αυτά βεβαίως είναι κοινό κτήμα, είναι, είναι δημοσιοποιημένα. Ελπίζω ότι σας απάντησα. Φων Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Νουή, επανέρχομαι στο Fiscal Backstop και το MREL. Από ό,τι έχω καταλάβει, η ιδέα ήταν να υπάρχει απέτηση bail-in, αρκετά γενναιόδορη όμως, σε σχέση με την ιστορική εμπειρία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όταν αυτό το μέτρο θα εφαρμοζόταν θα μπορούσε να υπάρχει ένα backstop στην περίπτωση όπου τα πράγματα πήγαιναν άσχημα. Και στην βάση του Μπέιλιν θα μπορούσε να στοχεύσει πλέον κανείς στο πρόβλημα ρευστότητα και όχι στο πρόβλημα της εξυγίανσης. Κάτι το οποίο, της καλύτερα, κάτι το οποίο θα διευκόλυνε εν τέλει. Εξεπλάγει λοιπόν όταν σας άκουσα να μας λέτε ότι το, οι απαιτήσει TLAC και MREL θα πρέπει να είναι σταθμισμένες στα διεθνή πρότυπα τη Συμφωνίας ΤΙΛΑΚ και όχι στα μέτρα που είναι απαραίτητα για το 8% του MRL που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Και επομένως το Ταμείο Διάσωσης Τραπεζών και ο μηχανισμός να μπορέσουν να δραστηριοποιούνται. Άρα πρέπει να στοχεύουμε περισσότερο στη Διεθνή Συμφωνία και με την EBRD στο κατόφλι των 7% είτε πρόκειται για μετοχικό κεφάλαιο είτε πρόκειται για δευτερεύον χρέος αυτή είναι η ερώτησή μου well, I did not say that it... δεν είπα ότι έτσι θα πρέπει να είναι λέγω μόνο ότι για τον πυλώνα 1 και 2 για τις απαιτήσει πυλώνος 1 και 2 για το κεφάλαιο. Είμαι βεβαία ότι αυτό που αναμένεται από εμά είναι να ζητούμε περισσότερο, περισσότερα από τις ε, πολύ μεγάλες διεθνείς τράπεζες και λιγότερα από τις μεσαίες και μικρές. Λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι είναι περίπλοκο. Αλλά αυτή είναι η απόφαση του ε, νομοθέτου. Είναι περίπλοκο να υπάρχει ευρωπαϊκό MR. L για όλες τις ε, τράπεζες. Γιατί θα είναι με μεγαλύτερη απέτηση από αυτό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο από τις παγκόσμιες ΣΥΦΙΣ. Συστημικές τράπεζες. Όχι. Συστημικές τράπεζες. Ναι. Το bail-in χαμηλώνει τώρα. Ώστε το bail-in του 8% των, ε, του χρέους εγώ δεν λέω των δανείων δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Αν όμως τα MREL διαμορφώνονται όπως το τιλάκ, άλλα δηλαδή κεφαλακά εργαλεία όπως κόκος και subordinated debt. E αυτό είναι διαφορετικό, διότι αυτό σημαίνει τότε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εκδίδουν πολύ την debt. E είναι... Και παρόλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο εξηγιάνσιμες τις τράπεζες διότι και πάλι το Μπέιλιν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που είναι εγγυημένες οι καταθέσεις. Uh, uh, Συγγνώμη για το μικρόφωνο. Θα μας ζητηθεί διαβούλευση έχω, έχω συζητήσει όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που αποφασίζει. Ούτε λέω ότι θα πρέπει να γίνει έτσι ή αλλιώς. Ο κ. Φουνβάτσεκερ, μια σύντομη συμπροματική ερώτηση. Διακόπτη πρόεδρο. Δεν άκουσα την ερώτηση. Σύμφωνα με τον νόμο, είναι μέλο του Μπεϊλίν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση και όπως είπαμε θα, συνεχίσουμε την συζήτησή μας όπως μας είπατε, μας θυμήσατε είμαστε συνομοθέτες και βεβαίω καλούμαστε να εφαρμόσουμε τους κανόνες που αποφασίζουμε είναι σωστό όμως και αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην ακρόαση. Πολύ σύντομα θα διεξαχθεί άλλη. Βλέπω εδώ ήδη τον Τζόναθαν Χιλ για το επόμενο πολύ, για την επόμενη πολύ σημαντική ακρόαση. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην δημόσια κρόση μα για την ε, τίτλοποίηση. Όπως βλέπετε έχουμε πολύ καλό πρόγραμμα και αναμένουμε και σημαντικές ε, συνεισφορέ για το νομοθετικό μας έργο. Όπως ξέρετε, Τώρα έχουμε σχέδια έκθεσης και για τα δύο σχέδια κανονισμών από τους εισηγητές μας όπως ξέρετε έχουμε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας και αναμένουμε τώρα βεβαίως τις τροπολογίες και το τελικό κείμενο για να ξεκινήσει και ο τριμερής διάλογος. να τελειώσει και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, Ένωσης ε, των Κεφάλαια Αγορών. Νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε με τον Τζόναθαν Χιλ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Βγάλετε. Θα κάνετε μια πρώτη τοποθέτηση και μετά θα ξεκινήσει η συζήτησή μας. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω και να σας μιλήσω για τις προτάσεις μας για να ξεκινήσουν ξανά οι αγορές της ε, τιτλοποίησης ε, και για να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό αυτό για να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ευρύτερη οικονομίας και να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τον κίνδυνο και για να παρουσιάσω το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε με έναν τρόπο συνετό μετρημένο που θα διδάσκεται και από το παρελθόν. Γνωρίζω πως η Επιτροπή έχει σκεφτεί πολύ το ζήτημα και γνωρίζω και τις εκθέσεις των κυρίων Τάγκ και Ζάλμπα για την πρόταση που έχουν κάνει και για τον κανονισμό κλοποίησης και τον κανονισμό κεφαλαϊκής επάρκειας. Αν πάρουμε ως αφετηρία την ε, κρίση πρέπει να θυμόμαστε πως τότε η τιτλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγαινε καλά και οι αμερικανικές τιτλοποίησεις δεν ανταποκρίθηκαν. Εμείς λοιπόν ενισχύσαμε το πλαίσιο διακυβέρνησης και διασφαλίσαμε την ορθή τους ε, ρύθμιση. Αυξήσαμε τις κεφαλιακές απαιτήσεις, εισαγάγουμε κανόνες για την συγκράτηση του κινδύνου για να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα. Αυξήσαμε την διαφάνεια τις απαιτήσει δέουσας επιμέλειας ε, θέσαμε ξεκάθαρες ε, προδιαγραφές ε, και αυξήσαμε την εποπτεία και τίποτα από αυτά δεν αμφισβητείται. Θεωρώ όμως πως τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες ερωτήσεις για να στηρίξουμε τις επενδύσεις για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι και να δούμε προσεκτικά τις αναλύσεις που δείχνουν τον θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τιτλοποίηση σε μια σύγχρονη οικονομία. Γιατί λοιπόν είναι σημαντική η τιτλοποίηση. Στην απλούστερη μορφή της η τιτλοποίηση μπορεί να είναι κάτι το απλό και να ωφελήσει ολόκληρη την οικονομία με το να μετατρέπει ατομικά δάνεια σε ομόλογα ανοίγουν οι επενδύσεις ε, σε, αγορα... σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μια πολύ ευρύτερη αγορά από τις τράπεζες. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα επιτρέπεται στις τράπεζες οι οποίες λαμβάνουν τις μηνιαίες πληρωμές από τα στεγαστικά δάνεια να τα συνδυάσουν αυτά τα δάνεια και να έχουν μια απόδοση για την επένδυσή τους. Έτσι μπορούν να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους, να μειώσουν το κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και να δανείσουν περισσότερο στην οικονομία. Έτσι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε επενδύσει που δεν θα είχαν αλλιώς και άμεσα οι ίδιοι. Η σημασία λοιπόν της τηλεοποίησης πηγαίνει πολύ πέρα από τον τομέα το χρηματοπιστωτικό. Ένας, μια αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί παραδείγματο χάρη να πουλήσει τα δάνεια τα οποία έχει δώσει για την αγορά αυτοκινήτων ένα πολυκατάστημα με, μια, με τις κάρτες τις οποίες έχει εκδώσει μπορεί με τον ίδιο τρόπο να αποκτήσει χρηματοδότηση. Μια εταιρεία η οποία μισθώνει εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να χρησιμοποιήσει την τίτλοποίηση ε, για να πουλήσει έτσι τις απαιτήσει που έχει για τις μελλοντικέ ε, πληρωμές για να αυξήσει τη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυξημένε πηγέ χρηματοδότησης και είναι ένα σημαντικό τρόπο για τις τράπεζες να διαχειριστούν κάποιον από τον κίνδυνο που πρέπει να αναλάβουν για να παρέχουν τι υπηρεσίε που χρειάζονται οι πελάτε του, όπω π.χ. στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. πω λειτουργεί αυτό. Κοιτάξτε, η τετλοποίηση είναι μια μεταφορά στοιχείων ενεργητικών όπως τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εκδοθούν κάποιοι τίτλοι και κάποια αξιόγραφα από τις ε, τράπεζες. Οι τράπεζες θα κρατάνε ένα μίνιμουμ 5% για να έχουν και αυτές κάποιο συμφέρον και τα υπόλοιπα μπορούν να απολυθούν σε θεσμικούς επενδυτές. Έτσι διαχέεται ο κίνδυνος, μειώνεται ο κίνδυνος σοκ και ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η τιτλοποίηση επίσης παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για τους επενδυτές, ειδικά τους θεσμικούς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες ή ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα σταθερής απόδοσης από τα καταναλωτικά και εταιρεικά δάνεια. Τα δε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά έχουν γνώση του κλάδου όπου χορηγούνται τα δάνεια. Οι θεσμικοί επενδυτές εκμεταλλεύονται αυτή την γνώση και χρησιμοποιούν την τιτλοποίηση για να έχουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προς όφελος των πελατών τους. Στο μακρό επίπεδο, η τιτλοποίηση μπορεί επίσης να στηρίξει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας σε ένα κοινό εγγραφό τους λένε πως το να φύγει κάποιο ποσοστό κινδύνου δανεισμού από τις τράπεζες θα είναι υποφελές για τις τράπεζες, για την ευρύτερη οικονομία και για την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμφωνούν και άλλοι μαζί τους. Νομίζω πως υπάρχει μια συνένεση μεταξύ των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών και των εταιριών που χρειάζονται τις ε, χρηματαγορές πως ισχυρότερα τέτοια μέσα τίτλοποίησης είναι επωφελή για την ευρωπαϊκή οικονομία και συμφωνώ και εγώ. Αυτή τη στιγμή η έκδοση τέτοιων προϊόντων στην Ευρώπη είναι χαμηλή έχει πέσει από τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε κάτω από 220 δισεκατομμύρια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στον κλάδο αυτόν έχει πέσει δε το επίπεδο της τηλεοποίησης στο κάτω από το μισό σε σχέση με την κατάσταση προκρίσης. Οπότε υπάρχουν λιγότερες επιλογές χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν και η πρότασή μας για να ξαναξεκινήσουμε την αγορά τυπλοποίησης καθορίζοντας απλούς και τυποποιημένους κανόνες. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή της ε, Βασιλείας και η ΑΕΟΣΚΑ. Βασιζόμαστε στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας Αγγλίας, ε, της Μικτής Επιτροπής και βεβαίως είχαμε και συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Προκύπτουν λοιπόν οι προτάσεις μας ε, από την ανάλυση ανεξάρτητων και σεβαστών ε, ιδρυμάτων. Βασίζομαστε λοιπόν σε προϊόντα τα οποία πήγαν καλά κατά τη διάρκεια της κρίσης και αποκλείσαμε αυτά τα οποία δεν λειτουργήσαν. Στόχος μας είναι να απελευθερωθεί περισσότερη πίστη στην ευρύτερη οικονομία, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία τιτλοποίησης η οποία θα πληρεί πολύ συγκεκριμένα κριτήρια απλότητας, ε, διαφάνειας και τυποποίησης με πολύ συγκεκριμένες κεφαλιακές απαιτήσει για όσους επενδύουν σε μια τέτοια τυπλοποίηση. Τι εννοούμε λοιπόν με απλότητα, ε, διαφάνεια και τυποποίηση. Απλότητα εννοούμε μόνο τυπλοποίηση η οποία θα έχει δάνεια συγκρίσιμα μεταξύ τους. Δηλαδή το να ανακατεύουμε καταναλωτικά με στεγαστικά δάνεια αποκλείεται. Εννοούμε την η οποία δεν ξαναπακετάρει άλλη προηγούμενη τυκλοποίηση και εννοούμε τυπλοποίηση όπου το προϊόν, το υποκείμενο δεν μπορούμε να το διαλέγουμε κατά πώς μας συμφέρει. Οπότε αποκλείονται εδώ πέρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για να διασφαλίσουμε ε, την διαφάνεια, αυτοί οι οποίοι θα πουλάνε τέτοια προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στους επενδυτές και στις ρυθμιστικές αρχές για να μπορούν αυτοί να κάνουν μια αξιολόγηση του κινδύνου και της απόδοσης και οι εξελίξεις στις σχετικές ευρωπαϊκές αγορές να παρακολουθούνται. Οι προτάσεις μας θα καταστήσουν υποχρεωτική την παροχή των σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά σε όλους τους επενδυτές και δωρεάν με τρόπο σαφή και συγκρίσιμο και για να υπάρχει η σωστή εποπτεία προτείνουμε ένα πλαίσιο βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εθνικών εποπτικών αρχών έτσι ώστε να ρέουν οι πληροφορίες και όλοι να τηρούν τους κανόνες. Γνωρίζω πως η Βερένα από την ΕΣΜΑ θα σας μιλήσει σε λίγο. Η ΕΣΜΑ θα παίξει ένα ρόλο όσον αφορά την ε, διαφάνεια του συνολικού πλαισίου. Τώρα, για την τυποποίηση. Στόχος μας είναι να δούμε τις τυποποίησεις εκείνες οι οποίες θα χρησιμοποιούν συνεπείς και κατανοητές δομές, όπου ο εκδότης θα διατηρεί και θα διακρατεί κάποιες από αυτές τις ε, τυποποίησεις και οι κανόνες θα είναι σαφείς εκ των προτέρων. Οτιδήποτε λοιπόν πηγαίνει σε μια τηλεοποίηση STS θα πρέπει να είναι αξιόχρεο σύμφωνα με τις ε, οδηγίες περί καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης. Εν ολίγης, τα κριτήρια για την τίτλοποίηση θα βοηθούν τους επενδυτές να αντιληφθούν σε τι επενδύουν. Έτσι, ο κίνδυνος των ε, υποκείμενων στοιχείων θα είναι πιο αντιληπτός και θα ενδυναμωθούν οι επενδυτές καθώς θα βασίζονται λιγότερο στην αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης και θα μπορούν μόνοι τους να κρίνουν βασιζόμενοι σε αξιόπιστα στοιχεία. Τα κριτήρια έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να διδαχτούμε από τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην Αμερικανική κατάσταση με τα subprime και να μην επαναληφθεί αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου τα διδάγματα της κρίσης. Πρέπει απλά όμως να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί, όχι να οδηγηθούμε σε αδράνεια και παράλυση. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ευρωπαϊκές τυπλοποιήσεις θα πήγαν πολύ καλύτερα από τις αμερικανικές. Οι τα χειρότερα προϊόντα 3α στην Ευρώπη ήταν 0,8% ε, το ποσοστό ε, χρεοκοπίας. Στην Αμερική ήταν 16% με τις γνωστές συνέπειες. Οπότε αυτό το οποίο λέω σήμερα είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μεν, αλλά να κοιτάμε και προς το μέλλον, να δούμε τις μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση και προτείνουμε μια έξυπνη λύση με βάση τις συμβουλές που λάβαμε από ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για να εκμεταλλευτούμε ως το δυνατόν περισσότερο τις ε, αγορές τιτλοποίησης της Ευρώπης έτσι ώστε να διοχετευτεί η χρηματοδότηση στην ευρύτερη οικονομία. Θεωρώ πως οι προτάσεις μας για απλές ε, διαφανείς και τυποποιημένε τυπλοποιήσει κάνουν ακριβώς αυτό. Ο Μάριο Ντράγκη είπε πως επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης αναβίωσης της αγοράς αυτής και της ανάγκης ενός προληπτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Υπάρχει λοιπόν ένα εύρωστο καθεστώς εποπτείας έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να λογοδοτούν μέσω ισχυρής εποπτείας και ταυτόχρονα παρέχουν μία αντιμετώπιση που σχετίζεται με τον κίνδυνο και ένα απλό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο για να επενδύσει κανείς σε ένα τέτοιο προϊόν. Γνωρίζουμε πως υπάρχει ένα κενό επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γνωρίζουμε πως οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερες ε, περισσότερα κονδύλια και θεωρώ πως η τυπλοποίηση η οποία θα είναι απλή, διαφανής και τυποποιημένη θα κάνει την διαφορά. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη απειλή στο μακρό επίπεδο την έλλειψη ανάπτυξης και ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε αυτές τις προτάσεις, να συμφωνήσουμε από αυτόν και με το να αυξήσουμε τις πηγές χρηματοδότησης να στηρίξουμε την ε, περαιτέρω ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Τζόναθαν για την εισαγωγική σας ε, τοποθέτηση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση και ολοκλήρωση της κρίσιμης αυτής νομοθεσίας. Θα αρχίσουμε τώρα με το πρώτο πάνελ μας. Καλώς ήρθατε Βερένα Ρος, διευθύντρια της ΕΣΜΑ και εσείς κύριε Γενικός Γραμματεύσης της Finance Watch, Finance Watch. Θα σας δώσω 7 λεπτά για τον καθένα. Τίτλος είναι «Διδαχθήκαμε κάτι από την χρηματοπιστωτική κρίση». Βεβαίω, θα είναι πολύ έντονα αλληλοσυνδεδεμένε τα δύο τμήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και τους εισηγητές για την τιτλοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκλησή τους έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον της τυπλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μιλώ ε, από πλευράς ε, ρυθμιστού αν θέλετε. Τρία είναι τα θέματα. Η σημασία μιας βιώσιμης και διαφανούς αγοράς τίτλων και η δεύτερον η δουλειά την οποία κάνουμε σαν έσμα ε, στα πλαίσια της τίτλοποίησης και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όπως επίσης και το θέμα της διαφάνειας έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τις σωστές πληροφορίες στα πλαίσια της τιτλοποίησης και είμαι στη διάθεσή σας πιθανώς για ερωτήσεις. Το θέμα του ρόλου τώρα της τιτλοποίησης στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ο Επίτροπος Χίλ τα είπε βέβαια, αλλά θα είμαι σύντομη. Όταν χρησιμοποιείται σωστά η τυπλοποίηση αυξάνει τη διαθεσιμότητα της πίστοσης και μειώνει το κόστος της χρηματοδότησης. Σαν μέσο χρηματοδότησης συνεισφέρει σε μια σωστή χρηματοδοτική βάση. Σαν μέσο μεταφοράς πιστώσεων μπορεί να βοηθήσει την αποτελεσματικότητα και την κατανομή των κινδύνων για την κάλυψη των αναγκών. Από την άλλη βέβαια όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά αναγνωρίζεται ότι η τιτλοποίηση λειτουργεί αποσταθεροποιητικά κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, μπορεί να εγκαταλειφθούν οι αγορές αυτές τιτλοποίησης αν δεν πιστεύουν οι επενδυτές ότι έχουν επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των κινδύνων ε, σχετικά με ένα συγκεκριμένο ε, προϊόν τιτλοποίησης και το κόστος του προϊόντος αυτό. Αυτό επίσης συμβαίνει όταν υπάρχει υπερβολική, αν θέλετε, λήψη υπόψη των αξιολογήσεων από πλευράς των εταιριών αξιολογήσεων, κάτι το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα τελευταία χρόνια εμείς σαν ΕΣΜΑ στον τομέα της τιτλοποίησης ρόλος μας βασικός ήταν να συνεισφέρουμε στην βελτίωση και την εφαρμογή του σωστού διακανονιτικού πλαισίου για να διασφαλίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη των αγορών τιτλοποίησης η εντολή μας μας οδηγεί στο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της τυπλοποίησης διατομεακά και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα σωστό ε, πεδίο, αν θέλετε, ανταγωνισμού και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Βασική μας, αν θέλετε, όμως ανησυχία είναι η προστασία ε, των επενδυτών. Να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές έχουν τις σωστές πληροφορίες και να κάνουν τις σωστές επιλογές. Όταν το πετυχαίνουμε αυτό, τότε θα έχουμε δημιουργήσει σωστές και σταθερές αγορές τυπλοποίησης. Σχετικά λοιπόν και με τη διαφάνεια η οποία απαιτείται για τους επενδυτές έχουμε αναπτύξει ε, και συγκεκριμένα τεχνικά μέσα τυποποίησης στα πλαίσια του κανονισμού CRA3. Κανονικά θα πρέπει να υπάρξει μια ιστοσελίδα από πλευρά τη ΕΣΜΑ όπου όλα τα εγγραφά θα μπορούν να είναι προσβάσιμα. Σχετικά τώρα με τη συνεκτικότητα της ε, οφειλόμενης αν θέλετε προσοχής και της δέουσας προσοχής έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα μέσα από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και από την ΕΙΟΠΑ και την ΕΣΜΑ ήδη από το Μάιο του 2015. Απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα, κοινή ορισμή και ένα συνολικό πλαίσιο επίβλεψης και εφαρμογής, επιβολής καλύτερα. Βασικό συμπέρασμα από τις προσπάθειες αυτές είναι ότι το θέμα μας είναι η διαφάνεια. Αυτό απαιτείται κυρίως για τους επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να έχουν πάρα πολύ σωστή πληροφόρηση για τις τιτλοποιήσεις και να μπορούν να τις συγκρίνουν. Έτσι λοιπόν ο κανονισμός που προτείνεται για την τιτλοποίηση, οι κοινοί κανόνες για τη δέουσα προσοχή και την διακράτηση και επίσης την ε, δημοσιοποίηση κανόνων για την τιτλοποίηση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε ε, την πληροφόρηση για τους επενδυτές διαθέσιμη. Αυτή είναι μια προσπάθεια στην οποία συγκεντρώνουμε την προσοχή μας. Οι συνομοθέτες στην Ευρώπη ήδη έχουν ε, πάρει μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας μέσω του CRA3. Υπάρχουν εκείνοι πίνακες και δημιουργήθηκε και μια ιστοσελίδα για τη δημοσίευση των πληροφοριών για τα λεγόμενα SFI, ε, τα διαθρωμένα ε, χρηματοδοτικά μέσα. Ε, αντιμετωπίσαμε βέβαια αρκετές δυσκολίες προσπαθώντας να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα SFI. Καταρχάς, τη απουσία μιας νομικής βάσης για τη συλλογή των τελών ή ενός χρηματοδοτικού φακέλου για την κάλυψη του σημαντικού κόστους δημιουργίας της ιστοσελίδας SFI. Αυτό μας δημιούργησε προβλήματα και σε μια πρώτη φάση ε, είδαμε ότι χρειάζονται αρκετά εκατομμύρια για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας. Υπήρξε πρόβλημα επίσης ε, για την εκχώρηση της δυνατότητας δημιουργίας του πίνακα SFI ε, σε, μια τρίτη πλευρά. Ε, παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τον κανόνα αυτό και τον πίνακα ο οποίος συνεπάγεται από τον κανόνα αυτό μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όπως είχε προβλεφθεί στα πλαίσια του CRA 3. Το θέμα είναι να δούμε τι είδους υποδομών θα στηρίξει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω ότι τα συστήματα για την παρακολούθηση των τιτλοποιήσεων και των δευτερευουσών στοιχείων ήδη υπάρχουν. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν νέες απαιτήσει για τις ιστοσελίδες των εκδοτών των τίτλων. Υπάρχει επίσης και το SFI και ο εισηγητής σας προτείνει επίσης, ο κ. Τάγκ, την δημιουργία ενός, ενός καταθετηρίου δεδομένων τυπλοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο έχει σημασία από τη δική μας πλευρά είναι αν οι επενδυτές θα έχουν ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τις ανάγκες τους και αν οι πληροφορίες αυτές θα διευκολύνουν τη δυνατότητά τους να συγκρίνουν και να επεξεργαστούν τα επίπεδα των δανείων και να δουν τις πιθανές διεξόδους ανάλυσης των κινδύνων και των αποδόσεων των τίτλων. Ε, όλες οι ε, πρωτοβουλίες λοιπόν για τη διαφάνεια θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο σωστής ε, διαχείρισης και να αποφύγουμε επικαλύψεις. Θα μπορέσουν λοιπόν οι επενδυτές να έχουν εύκολη πρόσβαση και κατανοητή πρόσβαση. Ε, οι πίνακες αναφοράς και η τεκμηρίωση είναι η βασική αν θέλετε, ε, πυρήνες αυτής της προσπάθειας ενημέρωσης. Η ΕΣΜΑ είναι έτοιμη λοιπόν να προχωρήσει σε τεχνικές ρυθμίσεις τυποποίησης ε, εφόσον μας δοθεί η εντολή. Θα χρειαστούμε για τα τεχνικά standards αρκετό χρόνο για να το κάνουμε σωστά και να διαβουλευτούμε σωστά με τους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 12 μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει να βοηθήσουμε όπου μπορούμε μέσω της τεχνικής μας εμπειρογνωμοσύνης. Είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστόφ, ευχαριστώ. Κύριο Σνάινταμ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο διότι η εμπειρία της Finance Watch μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε στην ερώτηση αν διδαχθήκαμε κάτι από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ο στόχος για τη δημιουργία της Finance Watch ήταν να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη φωνή δημοσίου συμφέροντος για να μπορέσει να αντισταθμίσει τα ε, ε, ιδιωτικά συμφέροντα που εκφράζονται στην χρηματοπιστωτική, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Με τους πόρους που διαθέτουμε προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε συζήτηση. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μέχρι τώρα πολλά έχουν λεχθεί για τις αιτίε και τις συνέπειες της κρίσης. Μία από τις συνέπειες ήταν ότι στο επίπεδο G20 αναλήφθηκε η υποχρέωση μεταρρυθμίσεων Κομισιόν και Κοινοβουλίο θα πρέπει να επενεθούν διότι κατάφεραν να προωθήσουν τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις για τη σταθεροποίηση του τομέα. Αυτό που είναι σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις από αυτές είναι microprudential. Το νόημά τους δηλαδή είναι να κάνουν να καταστήσουν ασφαλέστερα συγκεκριμένα ατομικά ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεν είναι του τύπου macro-prudential, ώστε να μπορέσουν δηλαδή να κάνουν ασφαλέστερο ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν λήφθησαν λοιπόν ορισμένα μέτρη, μέτρα, συγγνώμη, όπως το shadow banking. Ο βασικός στόχος του κανονισμού για, την, ε, για τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η σταθερότητα. Η μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δεν επέτυχαν να αντιμετωπίσουν την υπερβολική περιπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και άφησαν πολλές ευκαιρίες ανοιχτές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποφύγουν την ρύθμιση. Το CRD4 είναι καλό παράδειγμα. Δεν αφαιρέσαμε, δεν μπορέσαμε να αφαιρέσουμε τα υπερβολικά περίπλοκα εσωτερικά μοντέλα και τις ευκαιρίες για ρυθμιστικό arbitrage το οποίο συνεπάγονται. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο ε, ρωμαλαία Κάνουμε τώρα μια προσπάθεια αντισταθμίσεως βάζοντας ένα ακόμα επίπεδο περιπλοκότητας μέσω του bail-in. Η τιτλοποίηση και η κρίση θεωρήθηκαν ως αιτία και συνέπεια της κρίσης. Τώρα η τιτλοποίηση βρίσκεται στην καρδιά της νέας ατζέντα για την ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο πάνελ, τα περί Γι' αυτό έρχομαι περισσότερο στην ερώτηση αν συνάχθηκαν τα διδάγματα από την κρίση. Η απάντηση είναι καθαρά όχι. Όταν θα, φέρω σε, το, θα ρίξω το φως στην, στην θα σας εξηγήσω τι κάναμε πριν από την κρίση και τι κάνουμε τώρα. Πρώτα πριν από την κρίση δεν υπήρχε ευθυγράμμιση μεταξύ των αναγκών των ρυθμιστών και των επενδυτών. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν διαμορφώνονταν συγκεκριμένα κριτήρια Η στάθμιση του κινδύνου και το 5% δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να ανέλθει στο 20% το ποσοστό αυτό και περισσότερο και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια τομή μέσα από όλες από όλους, τους, από όλους τους κράτους. Το δεύτερο θέμα είναι η περιπλοκότητα των συναλλαγών που προκαλεί τελικά σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων φορέων. Το τρίτο θέμα είναι η υπερβολική εξάρτηση από τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας, αξιολόγηση δηλαδή της πιστοληπτικής ικανότητας. Τώρα, θα πρέπει πρώτα οι επενδυτές να ενθαρρυνθούν να ασκήσουν οι ίδιοι ε, την απαραίτητη δέουσα επιμέλεια και να μην αναμένουν από άλλους, δηλαδή από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τα κριτήρια STS, που να γίνεται από έναν φορέα που θα πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, για και έχει σημαντική ευθύνη απέναντι στους επενδυτές. Τέλος, το θέμα της συνθετικής ε, τυπλοποίησης. Συνεχίζεται η συζήτηση για το αν θα πρέπει να επιτραπεί μέσα στα πλαίσια του STS. Επιτρέψτε μου να επεκταθώ λίγο σε αυτό. Πολλοί πανεπιστημιακοί έδειξαν στη βάση εμπειρικών στοιχείων ότι η συνθετική τυτοποίηση αυξάνει τον το συστημικό κίνδυνο στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Και αναφέρω τα ονόματα Φράνκε και Κράνεν, Άλεν και Γκάλε και ούχτε και αλλά και αυτή η τελευταία το 2010. Όπως επίσης λένε τα Workstream, CBCBS και η OSCO, μόνο τυπτοποιήσεις πραγματικής κλίμακας ή σε μετρητών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να λάβουν την σήμανση STS βγάζοντας έτσι έξω από το πεδίο εφαρμογή τη συνθετική τυπλοποίηση. Αυτό συμβαδίζει και με αυτό που ε, ζητεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν δέχεται ως collateral τις συνθετικές τυπλοποίησεις. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, μελέτη δικτύπου που έκανε λέει καθαρά ότι η συνθετική τυπλοποίηση πρέπει να μείνει εκτός πλαισίου διότι είναι υπερβολική η περιπλοκότητα. Ανεξαρτήτως αν γίνεται για λόγους αρμπιτράζ ή μετρίασης του με η συζήτηση σχετικά με την συμπερίληψη ενδεχομένω τη συνθετική τυτοποίηση στο πλαίσιο STS πρέπει να σταματήσει. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τις αρχές βελτιωμένης νομοθεσίας και να χορηγήσει την κατάλληλη μελέτη αντικτύπου για να εξεταστεί η περαιτέρω ανάγκη, εάν υπάρχει, να ε, έχει διαφορετική μεταχείριση αυτού του είδους ιδιωτικοποίηση. Τώρα, έχουμε συναγάγει κάποια συμπεράσματα, η μνήμη μας όμως είναι πολύ σύντομη. Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η αποστολή. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμη και θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να έχουμε μια μειοπική αντιμετώπιση της αύξησης του καθάριστου προϊόντος σε βάρος της μελλοντική σταθερότητας. Θα πρέπει να αποφύγουμε να απορρίψουμε ως άσχετα τα επιχειρήματα των πανεπιστημιακών και να αγνοήσουμε τα επιχειρήματα φορέων που θα υποφεληθούν από το STS και που λένε ότι τούτη τη φορά τα πράγματα διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι η ορθή ρύθμιση είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η εντιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των οικονομιών. Κάτι το οποίο είναι μια αποστολή χωρί τέλο. Σα ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Γκουαρτιέρη, για την παρουσίαση του θέματο και θα δώσω το λόγο στου ευρωβουλευτέ. Με πρώτο τον Παύλο Σάλβα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστώ μάλλον και τον Επίτροπο Τζόναθαν Ιλ που έφυγε βέβαια στο μεταξύ. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, κεφαλαίες αγορές, χρειαζόμαστε βέβαια την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Πρόκειται και για βασική αρχή και ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγορές αυτέ πρέπει να είναι ανοιχτές και αποτελεσματικές έτσι ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη, να διευρύνουν την επενδυτική βάση όπως είπε και ο Επίτροπος και να διασφαλίσουν, προϋπόθεση μάλλον γι' αυτό είναι η σταθερότητα, η χρηματοοικονομική. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαίων όπως ακριβώς το προβλέπει στα πιστοτικά ιδρύματα και η Βασιλεία 2. Αυτό το οποίο με απασχολεί σε σχέση με το CRA είναι η, η ιεραρχία των αντιμετωπίσεων των ε, τρόπων με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Το ιδανικό θα ήταν οι τράπεζες να είναι από μόνες τους ικανές να χρησιμοποιήσουν τον πρώτο στη σειρά επί τη βάση των ε, ε, μοντέλων, των προτύπων που είναι υπό είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να είναι δύσκολο για διάφορους λόγους, σαν πρακτική. Η Βασιλεία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να υπάρξει μια πιο περιοριστική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτή που ακολουθήθηκε από το παρελθόν, στο παρελθόν και να διευκολύνουμε έτσι την χρήση της εσωτερικής μεθόδου. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι η άποψη των ομιλητών γύρω από αυτό. Και δεύτερον, σε σχέση τώρα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες των εκθέσεων και αναφέρθηκε λίγο σε αυτό στην αρχική του παρέμβαση ο κύριος Επίτροπος. Διαρωτώ με τι είδους πρωτοβουλίες μπορεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει ακόμα περισσότερο την τυπλοποίηση στο όνομα των μικρομεσαίων. Και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε και να συνεισφέρουμε με τις εκθέσεις αυτές στην δημιουργία νέων τρόπων χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι καλή αυτή η ακρόαση. Είναι πολύ καλό επίσης να δούμε α, ποια είναι τα μαθήματα της κρίσης τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν, της κρίσης που έχει προηγηθεί. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτική και η συζήτηση αυτή με τους πανελίστες είναι χρήσιμη. Το Κοινοβούλιο έχει ερωτήσεις πώς μπορούμε να είμαστε ικανοί σε προληπτικό επίπεδο, επιφυλακτικοί όσο χρειάζεται, να μάθουμε από τα μαθήματα του παρελθόντος, αλλά δεν είμαι βέβαια πεπισμένος ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κάνει αυτό πλήρως. Και γι' αυτό η ακρόαση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει. Να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις λοιπόν και να θέσω και κάποιες ερωτήσεις προς τους ομιλητές που προηγήθηκαν, ιδιαίτερα προς ε, την κυρία Ρώσ τη ΕΣΜΑ. Δύο ερωτήσεις για τη διαφάνεια πάντα. Η πρώτη. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις λέγουν ότι έχουμε μη ξεκάθαρα κριτήρια και μη ξεκάθαρες κυρώσεις για τον μη σεβασμό τους. Το να μην υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια αυτό δεν βοηθάει για την αναδημιουργία αυτής της αγοράς τυπλοποίηση, των αγορών μάλλον τιτλοποίησης. Κατανοείτε εσείς την κριτική αυτή από πλευράς των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών και πώς μπορείτε εσείς να καταστήσετε τα κριτήρια αυτά πιο ξεκάθαρα εξ αρχής. Δεύτερον, ε, να εμείνω λίγο στα θέματα της διαφάνειας Νομίζω ότι βασικό μάθημα από την κρίση είναι η ύπαρξη ε, έλλειψη μάλλον διαφάνειας ε, και για τους συμμετέχοντες στις αγορές, τους εμπλεκόμενους στις αγορές, αλλά και για τους επόπτες των αγορών αυτών. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε και αυτό το καταθετήριο. Ε, το θέμα είναι οι επενδυτές να έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση σε σχέση και με τα λεπτομερέστερα θέματα και όχι μόνο με τα κύρια χαρακτηριστικά και να δούμε ακριβώς τι επιθυμούν οι επενδυτές. Σε επίπεδο προληπτικό ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα ε, σε ποιο ε, επίπεδο θα σταματήσει η εξέλιξη του κινδύνου, γιατί θεωρητικά η τυκλοποίηση, βέβαια θα πρέπει να οδηγήσει στην ανακατανομή των κινδύνων και να καταστήσει τον χρηματοπιστό του μέσα αλλά αυτό μέχρι την πραγματικότητα έχει απόσταση. Για τον κύριο Νάινταμ, δεν ξέρω αν είναι γαλλικά, προφέρεται Νίνταμ, εγώ το λέω Ολλανδικά. Χαίρομαι που μας υπενθυμίσατε, χαίρομαι που μας υπενθυμίσατε ορισμένα στοιχεία σε αυτήν την ακρόαση κάποια στοιχεία τα οποία δεν καλύπτονται θα έλεγα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα οποία απαιτούνται βελτιώσεις. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τα περισσότερα από αυτά τα οποία αναφέρατε. Για να είμαστε όμως σίγουροι ε, είπατε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η λεγόμενη συνθετική τιτλοποίηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και τύποι όμως συνθετικής. Ε, εγώ καταλαβαίνω να αποκλείσουμε τα επικίνδυνα, αλλά όχι τις υγιείς μορφές συνθετικής, συνθετικής Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή όχι. Fox. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους δύο καλεσμένους μας. Οι ηγητές του ECR δεν είναι εδώ. Ο κύριος Καμάλ είναι ένορκος σε δίκη, αν το πιστεύετε. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή σε ένα δικαστήριο στο Λονδίνο. Γι' αυτό απουσιάζει. Συμφωνούμε λοιπόν πράγματι με την επιθυμία της Κομισιόν να αυξηθεί η τυπλοποίηση και ακούσαμε ενδιαφέρον τα νούμερα πως ε, τα ομόλογα 3α της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ένα ποσοστό 0,8% χρεοκοπίας ε, πριν την κρίση σε σχέση με το 16% των ΙΠΑ και αυτό τα λέει όλα. Να ρωτήσω λοιπόν, θεωρείτε πώς η αξιολόγηση και η στάθμιση του κινδύνου που γίνεται στην τιτλοποίηση στον τωρινό κανονισμό και σε σχέση με τον εγγενή κίνδυνο και σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης ε, μεταξύ των οποίων ε, και κρατικά και άλλα ομόλογα και γιατί για κάποιο λόγο φαίνεται ότι τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται ότι δεν έχουν κίνδυνο. Και έχω κι άλλο ένα ερώτημα και θα ήθελα ο κύριος Νίτζαμ να μας εξηγήσει εδώ πέρα. Εννοούσε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιος δημόσιος φορέας ε, που θα επιβλέπει τις κεφαλιακές απαιτήσει. Τι εννοεί, θα πρέπει να έχουμε ένα... μια υπηρεσία αξιολόγησης δημόσια. Για εξηγήστε μας τι εννοείται εδώ. Ευχαριστώ Μιχαήλ Τόιρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τους ε, πανελίστες εξ ονόματος ε, των Φιλελευθέρων ε, σε πρόσωπο των συνάδελφων τον κύριο Γκέζεκ ο οποίος απουσιάζει, γι' αυτό μιλάω αγγλικά. Γράφει λοιπόν για να προχωρήσουμε μετά την κρίση και να έχουν πρόσβαση μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην χρηματοδότηση. Η Finance Watch έχει επισημάνει πως αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ο Πέτερ και επίσης θα ήθελε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα εδώ πέρα γιατί σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση και υπάρχουν ακόμα κάποια μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Υπάρχουν βεβαίω οι ανάγκε ανάπτυξη και καινοτομία σε ένα περιβάλλον χαμηλή ανάπτυξη. Ε, και πιθανώς οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σήμερα να μην χρειάζονται ε, χρηματοδότηση από τις αγορέ, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει και να χρειαστούμε χρηματοδότηση για μια οικονομία η οποία θα αναπτύσσεται. Βεβαίω, οι τράπεζε έχουν το πρόβλημα ότι περιορίζονται από τι κεφαλαιακές απαιτήσει κάτι που είναι αναγκαίο δεδομένη της κρίση. Τι θα γίνει όταν θα έχουμε έναν κύκλο ανάπτυξης και θα θέλουν να επεκταθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συνεισφέρουν στην πραγματική οικονομία και επιπλέον η αγορά της τηλεοποίησης στην Ευρώπη έχει αποδειχθεί πολύ ασφαλέστερη από αυτή τον ΙΠΑ πρώτο 2007 επιπλεον Ο κ. Γέζα και επισημαίνει πως ανισχύει πάρα πολύ για το ποσοστό κατακράτησης 20% ε, του κινδύνου, κάτι το οποίο φοβάται ότι δεν θα επιτρέψει στο πλαίσιο αυτό του SDS να λειτουργήσει. Μήπως λοιπόν έτσι θα ενθαρρυνθούν οι χρήστες να πάνε σε άλλες αγορές όπως η Αμερικανική. Και έτσι θα δημιουργήσουμε ένα φρούριο Ευρώπη, κάτι το οποίο κατά την άποψη του Πετεργιζέκ δεν θα είναι σωστό για τις κεφαλαγορές ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, ε, ενώ θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική δεδομένου του έντονου παγκοσμίου ανταγωνισμού. Και τέλος, ο κύριος Γεζέκ θα έχει να αφαιρθεί στις ρήτρε περί τρίτων χωρών και το ερώτημα είναι προς την ΕΣΜΑ. Τι άποψη έχετε για τη θέση του Συμβουλίου και του εισηγητή για την διάταξη που λέει πως οι εκδότες θα πρέπει να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Και ε, υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τον Επίτροπο. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια του κυρίου Νίτζαμ για την ε, δύναμη του χρηματοπιστωτικού τομέα, γιατί συχνά ξεχνάμε την ε, κρίση αυτή και να τους δίνουμε όλο και περισσότερα περιθώρια. Και τελικά οι προτεραιότητες είναι του κλάδου και όχι όσων εκπροσωπούμε. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες πραγματικής οικονομίας και όχι του κλάδου. Και ίσως εδώ πέρα ακριβώς να μην βασιζόμαστε τόσο πολύ στις ανάγκες των ψηφοφόρων μας, αλλά στις ανάγκες των ενδιαμέσων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα λέω αυτά εισαγωγικά, γιατί θεωρώ πως είναι κίνδυνος για εμάς τους πολιτικούς το να μην θεωρείτε ότι ε, δρούμε προς το συμφέρον ε, των ψηφοφόρων μας. Και βλέπετε που οδηγεί αυτό στη χώρα μου. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, έχω κάποιες συγκεκριμένες ανησυχίες. Η πρώτη είναι από πού προέρχεται η ανάγκη για τιτλοποίηση και για το εάν θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προφανώς όλοι θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που ε, χρειάζονται, αλλά αν δείτε αυτές τις επιχειρήσεις και τις ρωτήσετε, ε, και την πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, μόλις 11% είπαν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. 25% είπαν ότι δεν έχουν πελάτες. Οπότε είναι περισσότερο οικονομικό το ζήτημα, ζήτημα λιτότητας ε, και την αποτυχία, την έλλειψη αγοραστικής δύναμης. Λοιπόν, για να έρθω στις συγκεκριμένες μου ερωτήσεις, για να επανέλθω στο θέμα της διακράτησης κινδύνου. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε βάρος στην διακράτηση κάποιου συμφέροντος των τραπεζών, έκθεση αν θέλετε σε μελλοντικό κείμενο, αλλά ε, τι θα λέγατε για την πρόταση να απαιτήσουμε από τις τράπεζες να διακρατούν τα δάνεια για λίγα χρόνια πριν τα ε, τιτλοποιήσουν για να μπορούν έτσι να έχουν κάποια ιστορικά στοιχεία για την διευθυντικότητα ε, τους. Μήπω θα μπορούσαμε έτσι να προτείνουμε έναν τρόπο μείωσης του κινδύνου ή ο κίνδυνος να παραμείνει συνδεδεμένος ε, με του εκδότες ε, των τίτλων. Πριν επιτρέψουμε να υπάρξει η τίτλοποίηση. Και η άλλη ερώτηση, γιατί θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπα Άσλη, για το ποιο θα κάνει την τίτλοποίηση. Και ποιο θα την πιστοποιεί. θα έχουμε μάλλον κάποια αυτοπιστοποίηση. Αυτό όμως ε, θα υπονομεύει την εμπιστοσύνη ή προτείνεται κάποιο δημόσιο φορέα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας από αυτό. Ευχαριστώ Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για κρίση η οποία ήταν στο παρελθόν, υπάρχει όμως ακόμα και τώρα. Ξεκίνησε από το 2008-2009 εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η κρίση αυτή, κατά κάποιο τρόπο, έγινε αντικείμενο σε εισαγωγικά εκμετάλλευσης για να υπάρξει ε, μια ρύθμιση του πιστοτικού συστήματος στην Ευρώπη, το οποίο αντί να συγκεντρώσει την προσοχή τους σε αυτό που προκάλεσε την κρίση, οδήγησε στη δημιουργία ενός πιστοτικού συστήματος, το οποίο βασίζεται σε παραδοσιακούς πάντα κανόνες, και δημιουργεί προβλήματα στο σύστημα αυτό. Και αναφέρομαι εδώ στις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν στα πλαίσια του Asset Quality Review, το οποίο θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον κίνδυνο στην πίστοση ενώ στα, σε πολύ πιο επικίνδυνα και θα έλεγα προβληματικά συστήματα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα. Νομίζω ότι όλο το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό, το πλαίσιο της βασιλείας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι το οποίο πιστεύετε λειτουργεί ικανοποιητικά ή απλά υποκύπτουμε στις ισχυρές πιέσεις των μεγάλων συστημικών τραπεζών προς ένα σύστημα διακανονισμού το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό και θα οδηγήσει σε περαιτέρω συστημικές κρίσεις. Θα πρέπει επίσης να πω ότι μιας και μέχρι τώρα δεν καταφέρνουμε εμείς να προχωρήσουμε σε μια σωστή διέρεση αν θέλετε του συστήματος του πιστοτικού το θέμα της ε, τίτλοποίησης θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση ορισμένων καρτέλ κάτι το οποίο όπως ακούγεται και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δεν είναι ικανοποιητικό. Και συμφωνώ με τις προτάσεις του Finance Watch, όταν λένε ότι σε σχέση με την παρουσίαση των νέων προϊόντων έτσι όπως προτείνονται οι διαδικασίες αυτές για τα νέα σύνθετα προϊόντα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και δεν μπορεί να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοιου είδους συστήματα και τέτοιου είδους προτάσεις για αγορά προϊόντων είναι ικανοποιητικοί. Το ίδιο σημαίνει επίσης και με τα συνθετικά προϊόντα. Είναι προϊόντα που εκμεταλλεύονται με καταχρηστικό τρόπο τα νομικά μέσα τα οποία υπάρχουν και δεν έχουν σχέση και δεν επηρεάζουν θετικά σε καμία περίπτωση την πραγματική οικονομία και δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα γιατί θα συνεχίσουν να λειτουργούν προβλήματα και σε κάποιες τράπεζες ενώ κάποιες άλλες θα κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα με τρόπο όχι σωστό. Η πραγματική οικονομία πάντως θα μένει απ' έξω και το πρόβλημά μας θα είναι συστημικό και η κρίση θα είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί εμείς με τα μέτρα μας θα μπορούσα να πει κανείς ότι γιγαντώνουμε το πρόβλημα που υπάρχει και αγνοούμε τους τρόπους λύσης του. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ποιος είναι ο κίνδυνος ο χρηματοδοτικός και όχι τόσο ο πιστοτικός. Ο πιστοτικός με κάποιο τρόπο ελέγχεται. Άνεμανς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ναι, ναι, ειδικά τον ε, κύριο με το ολλανδικό όνομα. Ναι, ναι, κοιτάξτε, η εντύπωση που αποκόμισα από τις διάφορες ε, προειδοποιήσεις ε, που ακούσαμε εδώ για την τυτοποίηση. Ε, όχι μόνο για την τιτλοποίηση βεβαίως, αλλά και για το τι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Ο Επίτροπος μίλησε για, μια, για ένα ευρωπαϊκό σύστημα τιτλοποίησης. Με κάνει να αναρωτιέμαι αν είναι απαραίτητο για αυτό το οποίο θέμε δουλειές και ανάπτυξη τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κινητοποιήσει την οικονομία, προχωράει σε νομισματική χαλάρωση. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία δηλαδή ενός ακόμα συστήματος. Η οικονομική προσθέμενη αξία. Γνωρίζουμε ήδη πως η τυπλοποίηση χρησιμοποιείται για να ενισχυθούν οι ισολογισμοί και έτσι τεχνητά να πούν κάποιοι ότι πληρούν τις προδιαγραφές της ε, βασιλείας, δηλαδή αφορά περισσότερο τον ίδιο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Δεύτερο ερώτημα γνωρίζουμε πως η τιτλοποίηση συνεισέφερε στην κρίση και οδήγησε ακριβώ ε, στο να μην υπάρχουν πλέον αυτές οι τοπικές ε, διαφορές ε, και είδαμε ακριβώ πως έγινε εξαγωγή του αμερικανικού προβλήματος στην Ευρώπη μέσω της Goldman Sachs. Ακόμα και εντός του ευρωπαϊκού συστήματος θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αυτές οι τοπικές ε, διαφορές. Κάτι το οποίο ήταν νομίζω μια αρκετά καλή προστασία για τις τράπεζες οι οποίες δρούσαν στην τοπική αγορά και ήταν απομονωμένες από το πρόβλημα στο παρελθόν. Τώρα όμως μέσω του ευρωπαϊκού αυτού συστήματο, δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η προστασία μέσω των περιφερειακών όπως είπαμε διαφορών. Και ίσως ενισχυθεί το πρόβλημα εντός ενός ευρωπαϊκού συστήματος ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος. Υπήρξαν πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να δώσω κάποιες απαντήσεις. Για το συνολικό πλαίσιο και για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να μπορέσει κανείς να κρίνει το τι είναι ασφαλές, το τι είναι σταθερό, τι είναι τυποποιημένο και τι είναι διαφανές. Απαιτούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και να περιλαμβάνονται επίσης και στη συγκεκριμένη αίτηση, αν θέλετε. Αυτό δεν είναι μόνο απλή δουλειά του EBA, αλλά πρέπει να υπάρξει κοινή ερμηνεία σε σχέση και με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και απαιτείται εδώ σύγκληση σε επίπεδο του λεγόμενου διακανονιστικού αμπιτράζου σε εθνικό επίπεδο. Απαιτείται λοιπόν και εδώ να υπάρξει μια δυνατότητα παρέμβαση ενδιαμέσου. Εδώ η ΕΣΜΑ θα μπορούσε να ε, καθορίσει τους μηχανισμούς αυτούς για να μην υπάρχουν κάποιες μορφές τυκλοποίησης που σε κάποια χώρα είναι νόμιμες και σε κάποια άλλη όχι. Το πιο σημαντικό στο οποίο αναφέρθηκα είναι η διαφάνεια για τους <clears throat> επενδυτές έτσι ώστε να κάνουν σωστές επιλογές. Αυτό δεν καλύπτει όμως την ανάγκη να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια επένδυση. Και αν αυτό μπορεί να επιδιωχθεί μέσω ενός συστήματος συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας κάποια από τα διαθέσιμα μέσα. Απάντηση γι' αυτό εγώ σήμερα δεν έχω. Για την στάθμιση του κινδύνων. Εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή. Είναι μια συζήτηση περισσότερο πρέπει να γίνει σε προληπτικό επίπεδο και όχι τόσο σε επίπεδο εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς. Για το τι προσπαθούμε να κάνουμε για να υπάρξουν πραγματικές ροές χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες. Βλέποντας επίσης το πρότυπο της χρηματοδότησης, προφανώς δεν μπορούν οι μικρομεσαίες από μόνες τους να προχωρήσουν σε τιτλοποιήσεις. Το θέμα είναι οι τράπεζες να μπορέσουν να τιτλοποιήσουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ενισχύοντας τον ισολογισμό τους να μπορέσουν να δανείσουν στις μικρομεσαίες καλύτερα και ευκολότερα. Το θέμα είναι λοιπόν η τράπεζα η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο βασικός αν θέλετε ε, παροχέας κεφαλαίων προς τις μικρομεσαίες να είναι σε θέση να το κάνει σωστά. Και άλλες δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το γιατί συγκεντρώνουμε την προσοχή μας ε, στα επιτρεπόμενα και προερχόμενα από την Ένωση προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε εμείς ε, τι δυνατότητες ελέγχου έχουμε σε επίπεδο νομοθετικό μπορούμε εμείς ε, να εντοπίσουμε ε, τους εκδότες που ε, βασίζονται, που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο και με την ίδια προσπάθεια να εντοπίσουμε τους επενδυτές. Νομίζω λοιπόν ότι οι ίδιοι επενδυτές μέσω ακριβώς της δέουσας προσοχής να γνωρίζουν αν μια τιτλοποίηση είναι δίκαιη, σωστή και τυποποιημένη. STS. Λοιπόν, είναι σαφές ότι απαιτείται να δούμε ένα σύστημα αναφορών, αυτό αναφοράς μάλλον, το οποίο έχει πλεονεκτήματα και είναι εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και μειονεκτήματα για το αν κάποιος εκδότης θεωρεί ότι το προϊόν του είναι προϊόν STS και σύμφωνα με ποια κριτήρια και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για την πιστοποίηση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται από επιχειρήσεις ή από αρχές οι οποίες να είναι με τη σειρά τους διακανονιζόμενες, ελεγχόμενες, να υπάρχουν κάποια κοινά επίπεδα τυποποίησης. Και αν είναι δημόσια υπηρεσία, τίθεται το θέμα αν θα είναι σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς μέσω της έγκρισης χαρτοφυλακίων, ή μέσω ευρωπαϊκού επίπεδου. Αν γίνει σε εθνικό επίπεδο, και επανέρχομαι σε αυτά που έλεγα, απαιτείται μια ιδιαίτερη σύγκληση των μηχανισμών εποπτείας των εθνικών έτσι ώστε να αποφύγουμε τις διαιτησίες. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας, λέει ο κύριος Νίνταμ. Θα προσπαθήσω πρώτα να απαντήσω σε κάτι που λέχθηκε και προηγουμένως και επανήλθε μετά στις ερωτήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή τίτλοποίηση. Ναι, απέδωσε καλά. Μόνο όμως σε ό,τι αφορά low to default rate. Όχι όμως για, για ε, τίτλους της τάξης, ε, με τιμές της τάξης του 8%. Εάν η αγορά, η ευρωπαϊκή αγορά τίτλοποίησης και μιλούμε για εμπορεύσιμους τίτλους, αν είχε λειτουργήσει καλά δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να αναζωογονοποιηθεί. Να ζαγωνηθεί, συγγνώμη. Για να χρειάζεται να την αναζωογονήσουμε πάει να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Υπάρχουν εμπορεύσιμοι τίτλοι, η αγορά τους όμως κατέρευσε με πρόκληση τεράστιων ζημιών στις, στους ισολογισμούς των επενδυτών, οι οποίοι έκαψαν τα χέρια τους. Και είπαν μετά, ε, εξ αμαρτήν ο καθόλου σοφού. Και εν τέλει, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πλαίσιο το οποίο θα ενσωματώσει τα διδάγματα του παρελθόντος. Και από την άποψη αυτή δεν νομίζουμε ότι η διαδικασία STS αποδίδει αυτή την αναγκαιότητα. Κατά την άποψή μας δεν είναι καθόλου απλή η διαδικασία αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των συνθετικών τίτλων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τους συνθετικούς τίτλους είναι να φύγουν από το ε, πλαίσιο STS, διότι δεν είναι απλοί τίτλοι, δεν είναι διαφανείς και δεν είναι τυποποιημένοι. Ναι, ε, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη ε, συνθετικών τίτλων, arbitrage και ισολογισμών, αλλά είναι δύσκολο καμιά φορά να διακρίνει κανεί ποιοι είναι οι υγιεί και ποιοι όχι. Μου ζητήσατε να επεκταθώ για τον ε, δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού. Κάτι είπε και σχετικά και η κυρία Ρένα Ρος, αλλά γιατί θέλουμε δημόσιο χαρακτήρα οργανισμό. Διότι γνωρίζουμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θα λειτουργήσει σωστά και μπορεί να ε, είναι και θύμα συγκρούσεων. Και η οίκη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι ιδιωτικέ επιχειρήσεις που βγάζουν μια πιστοποίηση τη πιστοληπτικής ικανότητα και είδαμε στο παρελθόν ότι δεν λειτουργεί αυτό. Και μιλούμε τώρα για το δημόσιο ε, συμφέρον και χρειάζεται λοιπόν ε, δημόσιους φορές. Εάν δούμε ότι δεν λειτουργεί αυτό θα θέλαμε και οι επενδυτές να ασκήσουν από μόνοι τους την δέωση επιμέλεια. Όσο όμως θα έχετε το λεγόμενο tranching, θα υπάρχουν κάποιες υποκείμενες επενδύσεις ή χρέη με ένα τριπλό β ή τριπλό σε που θα κυκλοφορούν στην αγορά. Και οι επενδυτές δεν θα κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν στην πραγματικά, δηλαδή να ασκήσουν την δέουσα επιμέλεια. Θα αγοράσουν τα χαρτιά αυτά θεωρώντας ότι κάποιοι έχουν ήδη ασκήσει την δέουσα επιμέλεια για λογαριασμό τους. Και θα κάνουμε το ίδιο λάθος με αυτό που κάναμε το 2007 και 2008, δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν εμπορεύσιμο τίτλο που υποτίθεται ότι είναι χαμηλά εμπορεύσιμος και αν αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα επειδή είναι εμπορεύσιμος τίτλος θα μπορεί να ξαναπουληθεί στη δευτερεύουσα αγορά. Εκεί όμως ισχύουν περίπλοκα εργαλεία και αυτό, το να, να υπάρξει εκεί αυτό το πράγμα είναι ψευδέστηση. Η ρευστότητα χάνεται, ε, χάθηκε διαμιάς στη διάρκεια της κρίσης. Υπάρχει το πρόβλημα λοιπόν αυτό του tranching και γι' αυτό ε, οι επενδυτές ε, δεν ασκούν την δέωση επιμέλεια που για μας είναι η λύση που προτιμούμε διότι εμείς θέλουμε οι επενδυτές να λειτουργήσουν πάλι ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές και όχι ως short term traders, δηλαδή να αγοράζουν και να πολλούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και βεβαίως η ε, έξοδος είναι πάντοτε πάρα πολύ μικρή για να βγει κανείς από τις διαδικασίες αυτές. Σε ό,τι αφορά τον αξιότιμο Γερμανό Ευρωβουλευτή που είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα credit supply. Εμείς θεωρούμε ότι για την ώρα ναι υπάρχει έλλειψη διάθεση από την πρώτη καταναλωτή. Και όταν εξετάζουμε την τιτροποίηση ή ε, ενώσει κεφαλαγορών σε σύγκριση με την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα στο παραδοσιακό γερμανικό σύστημα με τους ε, εγγύς φορείς όπως ε, τα ταμιευτήρια, ε, και τα κτλ. Έχουν πολύ καλά εξυπηρετήσει τις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μείζον πρόβλημα εκεί για το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα που χρηματοδοτεί άπαξ όταν έρχεται η ανάπτυξη αυτές τις μικρομεσαίες τουλάχιστον επιχειρήσεις στη Γερμανία. Συμφωνούμε με αυτά που λέχθηκαν για τις χρηματοπιστωτικές αγορές που είναι πολύ λιγότερο σταθερές από αυτό το proximity banking για ένα απλό λόγο. Η αγορά δεν έχει επενδυμένο συμφέρον στο, μέλος, στο μέλλον συγγνώμη, του δανειστού. Αν τα πράγματα πάνε καλά, ε, αγοράζουν τα πράγματα πάνε άσχημα, πολλό. Αυτά όμως οδήγησαν τελικώ στη συστημική κρίση. Και ποια είναι η οικονομική προστιθέμενη αξία του STS. Υπάρχει κάποια βεβαίως. Αλλά μόνο για τους ε, τραπεζικά εκείνα ιδρύματα που είναι πολύ μεγάλα για να τα αφήσουμε να ε, πτωχεύσουν. Όχι για τις άλλες τράπεζες. Η τιτλοποίηση του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ ήταν αποτυχία τελικά. Το να αναμένει κανείς ότι θα λειτουργήσει η τιτλοποίηση του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη εμένα με κάνει να διαρωτώ με μήπως είναι περισσότερο ευχολόγιο, γιατί έχουμε και τις 23 διαφορετικές γλώσσες, 28 διαφορετικά φορολογικά σύστηματα, 28 ε, διαφορετικές νομοθεσίες σχετικά με την πτώχευση. Ε, φανταστείτε τώρα, ισπανικά, ε, πορτογαλικά, ελληνικά, γερμανικά και το καθεξής. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στους επόμενους ομιλητές, τη δεύτερη μπορεί η τιτλοποίηση STS να αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Φάρκας. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από πλευράς της ε, εποπτικής μου αρχής, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να πάρουμε μέρος στη συζήτηση για την τιτλοποίηση, σημαντικό θέμα για ένα σωστό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα πρέπει να έλθει λοιπόν σε σχέση και με αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής να επανέλθει η ε, ταχαίως η εμπιστοσύνη. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των κεφάλαιων αγορών. Και η ευρωπαϊκή πρόταση και οι σφαιρικότερες παγκόσμιες προτάσεις από τη Βασιλεία βασίζονται στη σύσταση της ε, EBA του Ιουλίου 2015. Το STS, απλές διαφανείς και τυποποιημένες τυπλοποιήσεις, είναι ένα από τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εμπνεύσει τη Βασιλεία και την Αϊόσκο και θα εφαρμοστούν από ό,τι φαίνεται διεθνώς. Χαίρομαι λοιπόν που η EBA αποτελεί τον βασικό πυλώνα και της ευρωπαϊκής και της διεθνούς συνεργασίας. Η πρόταση τυπλοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του προηγούμενου φθινοπόρου είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και είναι υποδιαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι καλές οι προτάσεις αυτές, λειτουργούν σωστά προληπτικά και τεχνικά είναι σωστά διαρθρωμένα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία στοιχεία, τρία επιτεύγματα των προτάσεων αυτών. Πρώτον, καθορίζουν ε, μια νέα κατηγορία αγαθού το STS, σε επίπεδο τιτλοποίησης STS, κάτι το οποίο διασφαλίζει τυποποίηση και διαφάνεια που θα μειώσει ε, τους κινδύνους στην τιτλοποίηση που υπάρχουν όπως απέδειξε η κρίση. Αυτό στο κομμάτι το διακανονιστικό δεύτερον, οι προτάσεις αυξάνουν την ευαισθησία στους κινδύνους των απαιτήσεων των κεφαλαίων για τις τράπεζες και προτείνουν μια σωστή αντιμετώπιση έτσι ώστε να αναγνωριστεί το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου αυτού του είδους των συναλλαγών. Και τρίτον, βελτιώνουν τη συνεκτικότητα της νομοθεσίας ε, διατομιακά. Η τιτλοποίηση είναι σημαντικό θέμα για την EBA, την αρχή, την τραπεζική, γιατί αφορά φυσικά κυρίως ε, τραπεζικά προϊόντα. Οι τράπεζες είναι οι βασικοί παίκτες στην αγορά αυτή. Από αυτές προέρχονται τα προϊόντα της τιτλοποίησης και μαζί με άλλου τύπου επενδυτές θα έλεγα είναι, ε, παίζουν βασικό ρόλο. Η τιτλοποίηση επίσης είναι μέσο ε, πολλαπλασιασμού των τρόπων χρηματοδότησης και μεταφοράς του κινδύνου του πιστοτικού. Και τέλος, το βασικό στοιχείο του πλαισίου της τιτλοποίησης STS είναι μια σωστή προληπτική αντιμετώπιση της διαδικασίας δημιουργίας τους. Η δημιουργία ενός αυστηρού σετ κριτηρίων είναι, θα έλεγα, βασικό για τις προτάσεις τυπλοποίησης που διαχειρίζονται και προέρχονται από την τράπεζα. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχουμε εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της τυπλοποίησης και στα πλαίσια του συνθετικού πλαισίου και στα πλαίσια των παραδοσιακών δομών. Έχουμε δημοσιεύσει πρόσφατα τον Ιούλιο του 2015 την έκθεσή μας για την τυπλοποίηση STS, όπου είπαμε εμείς ποια είναι τα κριτήρια για τυπλοποίησεις υψηλής ποιότητας. Δημοσιεύσαμε επίσης το Δεκέμβριο του 2015 και την έκθεσή μας για συνθετικά προϊόντα τιτλοποίησης που δείχνουν ακριβώς την φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά των συνθετικών προϊόντων, ιδιαίτερα για συγκεκριμένα προϊόντα που βασίζονται από δάνεια μικρομεσαίων. Τρίτον, εμείς συλλέγουμε και ε, δημοσιοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια της διάθεσης κυκλοφορίας και κατάθεσης επίσης προτάσεων τιτλοποίησης, ε, όπως επίσης και τις κατευθυντήριες γραμμές, δημοσιεύσαμε κατευθυντήριες γραμμές ε, για θέματα μεταφοράς κινδύνων ε, μέσω της τιτλοποίησης τον Ιούλιο του 2014. Αυτό λοιπόν έγινε κατά τη διάρκεια και της νομοθετικής διαδικασίας που προηγήθηκε και που συνεχίζεται σήμερα. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις σε επίπεδο τίτλοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβάσαμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των εισηγητών της Επιτροπής σας την προηγούμενη εβδομάδα. Και γι' αυτό θα θέσουμε και τις δικές μας απόψεις σε κάποιες από τις δικές σας. Πρώτον, σχετικά το θέμα της ε, πιστοποίησης, αν θέλετε, συμμόρφωσης με τα κριτήρια STS. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη γενική αντιμετώπιση της πρότασης, ότι δηλαδή η βασική ευθύνη σε σχέση με τη συμμόρφωση προέρχεται από τους επενδυτές και από αυτούς από τους οποίους προήλθε το προϊόν. Νομίζουμε ότι οι προτάσεις ε, ε, που θα διασφαλίσουν την συνεκτικότητα των προτάσεων αυτών περιγράφονται σωστά. Τέτοιου είδους συμμόρφωση με τα κριτήρια STS λοιπόν είναι καλοδεχούμενη και δίδονται και τα μέσα για τη σωστή ερμηνεία ε, των κατευθυντηρίων γραμμών που περιλαμβάνονται στις προτάσεις. Σχετικά τώρα με τις συνθετικές τυπλοποίησεις, υποστηρίζουμε την εντολή της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής για μια έκθεση που θα οδηγήσει σε ένα πλαίσιο συνθετικών τυπλοποίησεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ πιο προσεκτικό τρόπο λόγω της περίπλοκης φύσης των προϊόντων. Οι τεχνικές μας προτάσεις σε σχέση με τις προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση του μηνός Δεκεμβρίου έγιναν δεκτές από την πρόταση την οποία κάνει η Επιτροπή σας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι ιδιώτες επενδυτές προστατεύουν την πίστοση ή παρέχουν προστασία στην πίστοση μέσω ε, μετρητών. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων για τις συνθετικές τυπλοποιήσεις STS. Τρίτον, σε σχέση με την κατακράτηση κινδύνων, παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι η πλειοψηφία των συστάσεων της EBA για την κατακράτηση κινδύνου, όπως περιλαμβάνονται στο έγγραφό μας του Δεκεμβρίου 2014, λαμβάνονται υπόψη από τους εισηγητές. Το 5% κατακράτησης, ε, το οποίο ε, απαιτείται από την πρόταση, είναι μια σωστή πρόταση η οποία θα επιτρέψει στους επενδυτές ε, να νιώσουν ασφάλεια και επιτρέπει επίσης και στους εκδότες να λειτουργήσουν με συμβατό τρόπο σε σχέση με το διακανονιστικό πλαίσιο. Αυξάνοντας τον κίνδυνο το ποσοστό αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως είναι σχετικά επικίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα σε μια προληπτική αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων και από την άλλη ε, πρόληψης των μη αναμενόμενων συνεπειών της λειτουργίας της αγοράς από την άλλη. Αν περάσουμε λοιπόν από το 5% σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό, σε οποιοδήποτε άλλο ποσοστό, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει υποχρεωτικά σε ένα βελτιωμένο επίπεδο συμπόρευσης, αν θέλετε, διαφορετικών συμφερόντων. Νομίζω λοιπόν ότι το πακέτο αυτό τιτλοποίησης είναι σημαντικό έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η αγορά τιτλοποίησεων. Σας ευχαριστώ για την πρότασή σας να σας μεταφέρω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Um, ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Γκάντι της Τράπεζας Σανταντέρ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας ομιλήσουμε για ένα θέμα που είναι σημαντικό για την πραγματική ευρωπαϊκή οικονομία. Η Σανταντέρ είναι από τους μεγαλύτερους εκδότες ε, τίτλων στην Ευρώπη μέσω του μητρικού ε, οργανισμού αλλά και των θηγατρικών είμαστε δραστήριοι σε 13 ε, ευρωπαϊκές χώρες και για ε, την πραγματικές, τις πραγματικές αγορές όπως υποθήκες, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιστοτικές κάρτες και έχουμε προσφέρει τα πλεονεκτήματα στην οικονομία. Λόγω της στατικής σημασίας της για μας ε, θεωρήσαμε και εμείς, ε, νιώσαμε και εμείς βαθύτατα δυσαρεστημένοι από την ε, κατάχρηση που έγινε στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποίησης που είχε αποδείξει την αξία της σε όλη την περίοδο της κρίσης τελικώς επλήγει ως αποτέλεσμα ενεργειών μεμονωμένων φορέων η ε, τιτλοποίηση είναι ένας βασικός πυλώνας των ευρωπαϊκών τραπεζών για να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τις ε, χρηματοδοτικές πηγές μαζί ε, με την συλλογή καταθέσεων, με καλυμμένα ομόλογα, με το χρέος και ούτω καθεξής. Μας βοηθεί επίσης να ανακυκλώνουμε το κεφάλαιό μας και να δανειοδοτούμε τους πελάτες μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό διότι η τιτλοποίηση είναι ε, από τις χρηματοδοτικές πηγές που ανέφερα προηγουμένως που επιτρέπει να ε, μοιραστεί κάποιους από τους κινδύνους των τυροποιημένων περιουσιακών στοιχείων με θεσμικούς επενδυτές δημιουργώντας έτσι τις ε, δυνατότητες να δοθούν ακόμα περισσότερα δάνεια ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν χρησιμοποιήσει και την πραγματική, το πραγματικό μορφότυπο πώληση αλλά και συνθετικούς μορφότυπους για τις ε, επενδύσεις αυτές. Έχουμε χρησιμοποιήσει την τιτλοποίηση για να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της στενότερης συμμετοχή στις κεφαλαίες για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Οι ε, επενδυτές μας λένε επίσης ότι εκτιμούν το εργαλείο της τιτλοποίησης διότι τους προσφέρει πρόσβαση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία πραγματικής οικονομίας χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να δαπανίσουν για τη δημιουργία ε, δαπανηρών υποδομών και τους προσφέρουν επενδυτικά προϊόντα που έχουν ε, χαμηλό συσχετισμό με τους ε, τραπεζικούς κινδύνους. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Santander και άλλοι φορείς που συμμετέχουν έχουν, παίξει σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση της ασφαλούς ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποίησης για να βοηθήσουμε τις τράπεζες να παίξουν τον ρόλο τους, να ενισχύσουν δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη και τους ε, στόχους της κεφαλαίου αγορά. Εμείς, καθώς και άλλοι φορείς που συμμετέχουμε, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε standards of excellence, βασισμένοι στις, βέλτι, στις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Χρησιμοποιούμε το, τη σφαγίδα ποιότητας PCS και θα συνεχίσουμε για να δίνουμε την ασφάλεια στους επενδυτές μας ότι αγοράζουν τίτλους ποιότητας. Έχουμε δημιουργήσει επίσης ένα shareholder και συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Δημιουργούμε μάλλον μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα καταθετήριο δεδομένων. Γιατί θέλουμε να υπάρχουν πληροφορίε ποιότητας ώστε οι να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Τέλος, συνεργαστήκαμε με άλλου συμμετέχοντε στον κλάδο για να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο στην σημαντική σας προσπάθεια να δημιουργηθούν κανόνες που θα αποφύγουν τις καταχρήσεις του παρελθόν και που κατέληξαν στο τρέχον πρόγραμμα STS. Μας ενθαρρύνουν οι προσπάθειές σας. Έχουμε λοιπόν συνεργαστεί με τους εταίρους μας στο AFME, EBF, EFR και άλλους για να προσφέρουμε επικοδομητικά σχόλια έτσι ώστε η STS να φτιαχτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σας απευθύνω έκκληση να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες και προτάσεις που έχουμε καταθέσει, ώστε η τελική μορφή του STS και το πακέτο CRR να μην τιμωρήσει άδικα τις πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλους ε, συμμετέχοντες που έχουν χρησιμοποιήσει ορθά το εργαλείο της τιτροποίησης. Για να αποφευθεί επιβάρυνση της αναζωογόνησης αυτού του σημαντικού εργαλείου για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος θα είναι ο κύριος Μέισμερ της ε, Landesbank της Βάδης Βιρτεμβέργης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές θα ήθελα να αναφερθώ στα πιθανά αποτελέσματα που έχει το προτινόμενο πλαίσιο τιτλοποίηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων χρησιμοποιώντα τα ABCP στην Ευρώπη. Τα ABCP χρησιμοποιούνται ω εργαλείο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, με πουλάνε τα προσδοκόμενα έσοδα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εκδίδοντας βραχυπρόθεσμα εμπορικά αξιόγραφα. Τα προσδοκόμενα έσοδα είναι κατά κανόνα αυτά τα οποία αναμένονται από τη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης ή από μισθώσεις ε, για να στηρίξουν την πώληση των τίτλων τους. Μπορεί να πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα ή οποιοδήποτε είδος αγαθών και υπηρεσιών. Σε πολλές περιπτώσεις ε, οι χρεωστέ ε, και όσοι μισθώνουν αυτές τι συναλλαγέ είναι μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Οπότε τέτοια προγράμματα με πολλαπλού ε, πολιτές είναι σημαντικό εργαλείο για την άμεση χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Όπως βλέπετε και στην ε, διαφάνεια, το ABCP με πολλού πολιτές είναι ένα χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό εργαλείο που έχει συσταθεί για να χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 80% των στοιχείων στα ευρωπαϊκά προγράμματα προκύπτουν από Ευρωπαίους πολιτές της πραγματικής οικονομίας. Και βεβαίως ε, η τράπεζα η οποία εκδίδει ένα τέτοιο πρόγραμμα, καλύπτει το πρόγραμμα και βεβαίως καλύπτει και όλους τους κινδύνους για τον επενδυτή. Τώρα, το εάν μια τέτοια συναλλαγή είναι απλή διαφανής και τυποποιημένη εξαρτάται από τις κεφαλαϊκές απαιτήσει ε, της ε, τράπεζας και άρα από το κόστος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Βλέπετε εδώ πέρα στη δεύτερη διαφάνεια πόσοι οι μέσες ε, συναλλαγές μίσθωσης θα έχουν μία αύξηση στη στάθμιση κινδύνου από 8-45% αν δεν είναι απλές διαφανείς και τυποποιημένες. Εάν είναι τυποποιημένες, παρόλα αυτά η στάθμιση κινδύνου θα τριπλασιαστεί. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα προσδεκόμενα έσοδα. Εδώ πέρα η στάθμιση κινδύνου θα μπορούσε να αυξηθεί από το 20% στο 60% για μία πλαίσια διαφανής και τυποποιημένες τυλοποίησης και μόνο στο 40% για τι ε, απλές διαφανείς και τυποποιημένε. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως το σχέδιο έκθεσης για την ε, τροποποίηση της οδηγία κεφαλαϊκή ε, επάρκεια απαγορεύει την χρήση της εξωτερικής αξιολόγησης. αυτού προτείνεται η τυποποιημένη προσέγγιση για όλες σχεδόν τις ε, ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, που θα εκδίδουν τέτοιους τίτλους σημαίνει πως η υφιστάμενη μεθοδολογία, η εσωτερική αξιολόγηση δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Κάποιοι πρώτοι υπολογισμοί έχουν δείξει πως η τυποποιημένη προσέγγιση θα οδηγήσει σε σαφώς υψηλότερες σταθμίσεις κινδύνου και άρα κόστος για την πραγματική οικονομία. Για να υπάρχει λοιπόν ένα αξιόπιστο και σταθερό μέσο χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία πρέπει να πετύχουμε τον ορισμό της απλής ε, διαφανής και τυποποιημένης τηλεοποίησης. Εάν οι ε, μηχανισμοί ρευστότητα για τις μέσες αυτές ε, συναλλαγές δεν είναι απλή διαφανής και τυποποιημένη, η αγορά απλά θα σταματήσει να υφίσταται. Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοια αρνητικά αποτελέσματα και στην αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης ε, που κυρίως χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουμε ακατάλληλους περιορισμούς όσον αφορά την λήξη των, στοιχείων, των υποκειμένων στοιχείων. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά βεβαίως έχουν στόχο να μην υπάρχει κάποια συνέπεια στην λήξη τους. Όμως αντιλαμβάνομαι πως επειδή η εκδίδουσα τράπεζα θα πρέπει να παρέχει πλήρη ε, κάλυψη ρευστότητας, ε, ήδη υπάρχει προστασία του επενδυτή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να υπάρχει σωστή και επαρκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει ο κανονισμό να σκεφτεί τον αντίκτυπο που θα έχει στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίων Τραπεζών έχει κάνει κάποιε προτάσει προσαρμογή του κανονισμού και βεβαίως θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε μαζί σας ε, λεπτομερώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ. Ίσως υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές ανάμεσα στον τρόπο που βλέπει ορισμένα θέματα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ιαν Μπέλ. Έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση. Όταν εμείς δημιουργηθήκαμε σαν μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, το ερώτημα που τέθηκε είναι υπάρχουν ασφαλείς τιτλοποιήσεις και αν ναι, τι μορφή έχουν. Σήμερα το ερώτημα αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το παρελθόν ξεκινήσαμε να δώσουμε μια, αν θέλετε, διανοητική απάντηση, όπως πιστεύουμε εμείς, με την αξιολόγηση των ζημιών των σοβαρών που προκάλεσαν κάποιες μορφές τυπλοποίησης το 7 και το 8. Ο ρόλος των subprime των Αμερικανικών και των λεγόμενων κύβων CDO ε, μας οδηγεί στο να δώσουμε απάντηση στην ερώτηση το τι είχαν αυτά τα προϊόντα τα οποία προκάλεσαν τόσο μεγάλη ζημιά. Η ίδια η τυπλοποίηση ήταν προβληματική. Τα προϊόντα που πρότεινε ήταν προβληματικά. Πώς ακριβώς θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο και πώς έγινε αυτό το οποίο έγινε. Μια λεπτομερής ανάλυση αυτών των καταστροφών, αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αυστραλία ή την Ιαπωνία, δείχνουν ότι κάποιες μορφές τυπλοποίησης δουλεύουν Αφεαυτής, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή μορφή τυπλοποίησης δεν είναι κάτι το επικίνδυνο και μπορεί να υπάρξει με ασφαλή τρόπο. Η ανάλυση την οποία κάνουμε και η οποία φαίνεται και στην εργασία ορισμένων δημοσίων οργανισμών όπως της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, δείχνει ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα που συνδυάστηκαν. Πρώτον, ε, το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διανομή αυτών των προϊόντων. Δεύτερον, η χρησιμοποίηση μαθηματικών προτύπων που στην ουσία ξεπέρασε τους αποδεκτούς, τις αποδεκτές παραμέτρους, η λεγόμενη ανατιτλοποίηση. Επίσης η εξάρτηση από την αναχρηματοδότηση των ιδίων των αγορών και όχι τόσο από την πληρωμή αυτών η οποία την επιστροφή την απόσβεση αυτών που είχαν δανειστεί τα συγκεκριμένα ποσά. Οδήγησαν όλα αυτά σε πάρα πολύ περίπλοκες καταστάσεις παντελώς ακατανόητες. Χωρίς την κατανόηση των αιτιών της κρίσης δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να αναζωογονήσουμε την αγορά τυπλοποίησης στην Ευρώπη. Το ερώτημα το οποίο τίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα είναι αν η πρόταση STS έχει μάθει από τα μαθήματα του παρελθόντος. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της πρότασης αυτής που πράγματι καλύπτουν αυτά τα προβλήματα τα οποία εντόπισα προηγουμένως και τα οποία πιστεύουμε ότι βρίσκονται στη ρίζα των προβλημάτων του 2008. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση μπορεί να αναζωογονήσει την αγορά. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία σκεπτικισμού. Κάποια στοιχεία επίσης ε, και για το τι λείπει στην πρόταση. Καταρχάς υπάρχουν κάποια στοιχεία μηχανισμών αγοράς που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να επενδύσουν ασφαλώς. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις εκθέσεις ε, του Κοινοβουλίου σχετικά με τους επενδυτές ε, να προχωρήσουν στη λεγόμενη ε, οφειλόμενη ιδέουσα επιμέλεια αν θέλετε ή προσοχή για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους και να κάνουν τη βασική δουλειά που απαιτείται από αυτός. Επίσης οι εκδότες θα πρέπει να είναι πλήρως ε, υπόλογοι για τις πληροφορίες τις οποίες ε, δημοσιοποιούν. Συμφωνούμε με αυτά τα δύο. Όμως πιστεύουμε ότι ε, μια θεμητή διαδικασία από πλευράς της κοινότητας των επενδυτών είναι να υπάρχει ένας μηχανισμός πιστοποίησης που να τους βοηθά να κάνουν σωστά ε, τον έλεγχο των μηχανισμών συμμόρφωσης, διαφορετικό από τον έλεγχο που θα κάνουν οι ίδιοι. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω ορκωτών λογιστών ή μέσω, αν θέλετε, ε, των στοιχείων που παρέχει το MIFID, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη σωστή ανάλυση. Σημειώνουμε επίσης και την αναφορά της έκθεσης σε ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερμηνείας. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, αυτό είναι θετικό και παρατηρούμε επίσης και την έκθεση της έκκλησης για ένα είδος καταθετηρίου έτσι ώστε να διατηρούνται όλα τα στοιχεία και νομίζω οι επενδυτές κάτι τέτοιο θα το καλοδεχθούν. Είμαι στη διάθεσή σας για να δώσω περαιτέρω απαντήσεις. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάμπορ είναι η τελευταία ομιλήτρια από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας, στο Μπρίστολ. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γκαμπόρ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση. Μα ζητήσατε να δώσουμε την απάντηση. Μπορεί η τιτλοποίηση STS να αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Δύο σημεία. Πρώτον, αν χρησιμοποιούμε τη δημόσια παρέμβαση για να δώσουμε ανάσα στις αγορές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Σε επίπεδο προσφοράς λέγεται ότι η τιτλοποίηση θα βοηθήσει την πρόσβαση των αγορών στην χρηματοδότηση και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Γνωρίζουμε όμως ότι οι μικρομεσαίες ανησυχούν περισσότερο για να βρουν πελάτες παρά για τη χρηματοδότησή τους. Έχουμε στοιχεία επίσης ότι οι μικρομεσαίες λειτουργούν καλύτερα σε χώρες με μεγάλους αριθμούς τραπεζών, πιστοτικών ιδρυμάτων, όπως τα μιευτήρια, συνεταιριστικές τράπεζες κτλ. Συνεπώς εκεί βέβαια θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση όπως και στο παρελθόν. Αν τα μαθήματα του παρελθόντος βοηθούν, τότε άλλοι τύποι δανειστών σε σχέση ε, με την αγορά κατοικιών αν θέλετε ή αγαθών διαρκείας, τότε εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποια νέα στοιχεία. Αλλά αυτό μερικές φορές ε, οδηγεί και στην δημιουργία ε, φούσκας σε εισαγωγικά στον τομέα της αγοράς κατοικίας. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά εμπόδια λοιπόν στο συνδυασμό των δανείων τη στιγμή που ένα γερμανικό δάνειο σε μικρομεσαία και ένα ελληνικό δάνειο σε μικρομεσαία έχουν το ίδιο μέσο τυπλοποίησης είναι κάτι το οποίο προς το παρόν φαίνεται πολύ μα πολύ μακρινό. Μπορεί να μην έχει σημασία το ότι ε, τα STS όταν είναι σωστά σχεδιασμένα θα αναζωογονήσουν τους εθνικούς, τις εθνικές αγορές τίτλοποίησης και όχι τόσο τις ευρωπαϊκές αγορές. Εδώ θα βρούμε αν θέλετε κάποιες επιπτώσεις και από το CMU. Το CMU, η πράσινη βίβλος, μαζί με το έγγραφο της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέει ότι υπάρχει θεσμική ζήτηση για τέτοιου είδους assets η εμπλοκή των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιριών είναι κάτι το οποίο μέσω της στρατηγικής αγοράς για, παρακράτη, για κατακράτηση είναι κάτι που θα βοηθήσει τις αγορές τυπλοποίησης. Η οικονομική θεωρία όμως και η εμπορία από τις προηγούμενες κρίσεις μας μαθαίνουν να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα σε ρευστές αγορές. Αυτή ήταν και η θέση της ΑΦΜΕ, της Ένωσης Χρηματαγορών της Ευρώπης μετά από τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου. Η πτυτικότητα των τιμών είναι υψηλή σε εμμύρευστες αγορές και αυτό θα φανεί στους ισολογισμούς των επενδυτών γιατί οι κανόνες συλλογιστικοί απαιτούν τη δημοσίευση της αξίας των δανείων σε τιμές αγοράς. Βλέποντας το τι έγινε το 2007 με 2008, αυτό οφείλεται ε, στη λεγόμενη διαδικασία mark to market. Ε, γι' αυτό ακριβώς η έρευνα από πλευράς της ε, Τράπεζας της Αγγλίας οδήγησε στο ότι οι λογιστικοί κανόνες δίνουν κίνητρα στις εταιρείες να αγοράζουν όταν είναι ψηλές οι τιμές και να πολλούν όταν είναι χαμηλές. Η ρευστότητα της αγοράς είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβει κανείς. Ακόμα και η αμερικανική αγορά ομολόγων πρέπει να σέβεται 55 κριτήρια για να μπορέσει κανείς να ταξινομήσει τα προϊόντα αυτά στα πλαίσια της ετικέτας STS. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχει να λάβει μια πολύ σημαντική απόφαση σε ένα πολύ τεχνικό θέμα. Αλλά σε επίπεδο πολιτικό είναι απλό το θέμα. Όταν ψηφίσετε για τα κριτήρια του STS, ψηφίζετε για το δημόσιο δίκτυο ασφαλείας το οποίο θέλει να βρίσκεται κάτω, πρέπει να βρίσκεται κάτω από τις ε, τιτλοποιήσεις στην Ευρώπη. Τα κράτη δεν μπορούν να αφήσουν να αυξηθεί το κοινωνικό κόστος των δανειοδοτήσεων των ε, ιδιωτικών συντάξεων. Η ερμηνεία, η ευρύτερη του τι εννοούμε εμείς ε, με τον όρο STS θα βοηθήσει να έχουμε πιο, αγνά προϊόντα θέλετε, μικρότερη περιπλοκότητα και μεγαλύτερη εμπλοκή και γνώση όλων των συμμετεχόντων σε αυτές τις αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είχαμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ο Ζάλμπα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου μου Ότμαρ Κάρας. Το... θέμα αυτό της ε, τιτλοποίησης είναι ένα σημαντικό εργαλείο και για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και για την πραγματική οικονομία. Σε σύγκριση με τις ΣΥΠΑ πρέπει να πούμε πως οι ευρωπαϊκές τιτλοποιήσεις τα πήγαν πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ε, οι ευρωπαϊκές τιτλοποιήσεις 3α ε, είδαν ένα πάρα πολύ χαμηλότερο ποσοστό μη σε σχέση με τα αμερικανικά αντίστοιχα. Ο στόχος ε, της νομοθεσίας αυτής είναι άρα να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στα μέσα αυτά. Στόχος μας πρέπει να είναι να υπάρξει αυτή η τιτλοποίηση ως ε, ένα ελκυστικό επενδυτικό προϊόν. Εάν επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία και να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Οι διαχειριστές ε, επενδύσεων ε, θα πρέπει βεβαίω να, κάνουν, να ασκούν τη δέωση επιμέλεια για τους πελάτες τους. Πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι ευθύνες και να αναλυφθούν κάποιες δράσεις για να προληφθούν ε, εγκληματικές ενέργειες. Αλλά βεβαίως οι αυστηρές απαιτήσει για αστική ευθύνη σημαίνει πως ίσως υπάρχει ένα κίνδυνος τον οποίο κάποιοι δεν θα ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν. Και βεβαίως όλα αυτά θα έχουν ε, την συνέπεια της αποτροπής επενδύσεων στις δηλοποίησεις σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων. Θα μπορούσε μια ανεξάρτητη πιστοποίηση από τρίτους να δικαιολογήσει την πλήρωση των κριτηρίων για πλήρη διάφανη και τυποποιημένη τυλοποίηση. και θα μπορούσε έτσι να έχει μια διασφάλιση ο επενδυτής. Τι μορφή θα μπορούσαν αυτά να πάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει το κείμενο αυτή τη στιγμή, μόνο οι επενδυτικές εταιρείες έχουν ε, την δυνατότητα και μάλιστα όσες είναι επιστοποιημένες σύμφωνα με την MIFID να αναλάβουν τέτοια ε, έργα τετλοποίησης. Είναι σωστό αυτό ή πώς θα έπρεπε να διερευνήσουμε την δυνατότητα να δούμε και τα ταμεία τα οποία είναι επιστοποιημένα σύμφωνα με την οδηγία usage Είναι θετικό το ότι αυτό έχει περιληφθεί στην πρόταση της Κομισιόν. Κατά την άποψη της ε, Κομισιόν του Συμβουλίου και άλλων ε, θεωρείται πως ε, με μια πιο αυστηρή ρύθμιση θα ευνοηθούν περισσότερο εκείνοι οι τίτλοι με πιο μακροπρόθεσμη λήξη. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να εξορροπηθεί ο κίνδυνος και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω την αποψή σα ε, για αυτό το οποίο προτείνει ο συγητή για την διακράτηση κινδύνου. Στόχος λοιπόν εδώ πέρα είναι να υπάρξει μια διάχυση του κινδύνου. Η αύξηση λοιπόν του ωρίου από το... Η μείωση του από το 20% στο 5% φαίνεται πώ είναι αντίθετη με αυτόν τον στόχο. Μπορείτε λοιπόν να μα πείτε ποιε είναι οι απόψει σα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φενάντες, ευχαριστώ πολύ. Και πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πρόσωπα που συμμετέσχουν στο πάνελ και για την προπαρασκευή και για τις τοποθετήσεις τους. Ακούσαμε τα διάφορα επιχειρήματα σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα τα που έχουν ε, προκληθεί και ότι δεν είχαν τόσο πολύ σχέση με την προσφορά όσο με την ζήτηση και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είχαν, ε, είχαν ε, πρόσβαση σε πιστώσεις. Τα, οι παραδοσιακές πιστώσεις εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, όμως ένα μέρος του προβλήματος της ζητήσεως ασφαλώς έχει κάποια σχέση και με την δυσκολία που βλέπουμε στην χρηματική πολιτική και την εφαρμογή της, την νομισματική πολιτική. Ε, το πρόβλημα αυτό, μάλλον να το πω διαφορετικά, το σύστημα αυτό των τιτλοποιήσεων έχει ως στόχο να εφαρμοστεί μια πολιτική χρήματος, δηλαδή να ενισχυθεί η ζήτηση, κάτι το οποίο θα ωφελήσει όλη την οικονομία. Από τις διάφορες τοποθετήσεις Άκουσα να θίγονται κάποια βασικά θέματα που είναι σημαντικά και για την έκθεση. Βέβαια δεν μιλήσατε όλοι και όλες για όλα τα θέματα που μας, μας απασχολούν. Στην έκθεση ΤΑΝΚ προτείνεται να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων για τους επενδυτές. Θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχετε. Αυτό θα ήταν μια προσπάθεια, δηλαδή αύξηση της διαφάνειας του συστήματος ΕΣΤΕΣ. Επίσης, ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ της αύξησης του ποσοστού από 5% σε 20%. Ακούσαμε βέβαια και τα αντίθετα επιχειρήματα. Επίσης, το... ποια είναι η άποψή σας. Επίσης, το πρόβλημα της πιστοποίησης. Εδώ χρειάζεται ένα σύστημα που να είναι απολύτως διαφανές. Άλλο ερώτημα που απασχόλησε και τον κύριο Ζάλμπα. Τι γίνεται με την ιεράρχηση των συστημάτων υπολογισμού των κεφαλακών απαιτήσεων. Και αυτό ισχύει και για τη ρύθμιση. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ. Thank you. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά παρακαλώ. Οπλιστείτε με τα ακουστικά σας. Κατά βάση να αντιμετωπίζουμε πολύ θετικά την πρόταση STS που θεωρούμε ότι είναι καλός τρόπος για να ξαναπάρει μπρος η τιτλοποίηση. Βέβαια, δεν είναι μονάχα η ανάγκη δημιουργίας του STS ως εργαλείου, αλλά να βρεθεί και η σωστή ισορροπία σε ό,τι αφορά τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Είδαμε λοιπόν ότι όταν σταθμίζονται οι κρατικοί τίτλοι με μηδέν, ενώ οι τίτλοι της ε, με υψηλά ποσά δεν λειτουργεί το σύστημα και στεγνώνει η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να ενισχυθεί η αγορά της τιτλοποίησης όταν αυξάνοντας δηλαδή και τη στάθμιση των ε, κρατικών τίτλων. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την μείωση των απαιτήσεων, κεφαλαϊκών απαιτήσεων του STS, τι συνέπεια θα έχει στις τιτλοποιήσεις που ε, δεν επωφελούνται από αυτό, διότι είναι δυνατόν να γίνει ε, εκεί. Για παράδειγμα, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μήπως εκεί προκληθεί νέα έλλειψη ισορροπίας, ώστε η τιτλοποιήσιμες απαιτήσει στα πλαίσια του STS τελικά εποφεληθούν περισσότερο οδηγώντας έτσι σε μια έλλειψη ισορροπίας απέναντι σε εκείνες οι οποίες δεν μπορούν να τιτλοποιηθούν στα πλαίσια του STS. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Τόιρερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς, οι φιλελεύθεροι, υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, δημιουργία του STS. Ευχαριστούμε δε ιδίως τον ε, Πρόεδρο για την επιλογή των πάνελιστ. Βέβαια, μας προκαλεί κάποιες ανησυχίες η, ε, τα αποτελέσματα της ακροασούς σε ό,τι αφορά τα commercial papers. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις, ιδίως για τα ABCP, Asset Backed Commercial Papers για, να μπορέσουν λοιπόν να βελτιωθούν οι δυνατότητες της α, ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποίησης χρειάζεται ταχεία προώθηση των δύο νομοθετικών σχεδίων και εμείς δεν θέλουμε να συνδυαστούν με τις διαβουλεύσεις για το έντις. Τώρα, ε, έχω μια ερώτηση για τον ο Μέισμερ. Αν κατάλαβα καλά, φοβήστε ότι τα ABCP στο μέλλον δεν θα είναι, δεν θα είναι πλέον δυνατά. Ε, θα είναι δηλαδή εφικτά με το επιχείρημα ότι η βασική προσέγγιση είναι υπερβολικά δαπανηρή. Και αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, είναι ότι η internal rate based approach βασίζεται και στο external rating. Μήπως μπορείτε να εξηγήσετε περισσότερο τι εννοείτε. Και μια, ε, δεύτερη, ε, ένα δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι η απέτηση ότι οι originator και οι, μελλοντικοί, και οι, και οι, και οι original lenders μπορεί και ο συνδυασμός αυτός να οδηγήσει στο μέλλον ABCP να μην είναι πλέον εφικτά. Εγώ δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των ε, σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για την πραγματική οικονομία ναι, πλέον, να μην είναι πλέον δυνατά αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό απευθύνω ερώτηση και στην Κομισιόν συμφωνεί ότι όντως πρέπει να υπάρχει ανησυχία σχετικά με το ότι μπορεί να μην είναι διαθέσιμα πλέον στην πραγματική οικονομία τα EBCP και ποιε θα είναι οι συνέπειες στην ε, ευρωπαϊκή αγορά ότι για παράδειγμα πωλήσει αυτοκινήτων δεν θα μπορούν πλέον να τυπλοποιούνται ούτε leasing μηχανημάτων για παράδειγμα και κάτι τέτοιο θα σήμαινε μια ε, βαρύτατη απειλή ε, σε βάρος της μελλοντικής ευρωπαϊκής οικονομίας ευχαριστώ, Μίγκελ Βιέγκα. Ευχαριστώ γρήγορα, γιατί βλέπω πως έχει περάσει η ώρα. Αυτά τα προϊόντα ήταν ε, στις ρίζες ε, της ε, οικονομικής κρίσης. Και αν δούμε αυτό το σχέδιο κανονισμού δεν μπορώ να πω πως αυτά τα προϊόντα είναι ούτε απλά ούτε διάφανα. Και δεν με έχετε πείσει. Και μάλιστα η συζήτηση αυτή δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η όλη διαδικασία. Είχαμε κάποιες σοβαρές αμφιβολίες για την υποπτία του συστήματος ε, στο σύνολό του και νομίζω πως ε, έχουμε σοβαρούς λόγους. Ανησυχούμε για τις δυνατότητες εποπτείας αυτών των προϊόντων στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί τα περισσότερα δάνεια που μετά τιτλοποιούνται το μιλάμε για κίνητα είτε για φοιτητικά δάνεια κτλ. Οι πηγέ τους είναι τέτοιες. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Ε, τι συνέπεια θα είχε η απαγόρευση αυτών των προϊόντων. Εντάξει, οι τράπεζες θα έπρεπε να κρατήσουν τα δάνεια αυτά στον ισολογισμό τους. Και αντιλαμβάνομαι πως αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τιτλοποίησης, αλλά πέρα από την δυνατότητα των τραπεζών να ξεκαθαρίσουν τα... τον ισολογισμό τους. Τι συνέπειες έχουν αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Σκοτ Κέιτο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να καλωσορίσω και τον συνάδελφο που είναι από τον Πρίστολ. Έχω δύο σοβαρά θέματα εδώ. Το πρώτο αφορά όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε αυτά τα στοιχεία του ισολογισμού των τραπεζών. Αλλά αν πάνε σε άλλους ισολογισμούς τραπεζών στο πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος, ποιο είναι το όφελος. Γιατί νομίζω μάθαμε από την κρίση πως οι τράπεζες είναι διασυνδεδεμένες και απλά ο ένας πάσαρε τον κίνδυνο στον άλλον. Οπότε ποιο είναι το όριο το οποίο εσείς θα προτείνατε για να είναι οι τράπεζες και επενδυτές πέρα από εκδότες. Το δεύτερο ερώτημα είναι κάπως πρακτικό. Είναι το ποιος θα επιτρέπεται να τα εκτίδει αυτά τα προϊόντα. Οπότε θα ήθελα εγώ να προτείνω την ιδέα ειδικευμένων οίκων τιτλοποίησης που θα είναι πιο αποτελεσματικοί, θα έχουν ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς όσον αφορά και την έκδοση και την αποθήκευση των προϊόντων αυτών και θα είναι οχήματα ειδικού σκοπού και μόνο από εκεί θα μπορεί κανείς να αγοράζει τέτοια προϊόντα. Η μία πλευρά είναι αυτή και η άλλη πλευρά είναι η πιστοποίηση αυτών των προϊόντων. Και πάλι εδώ θα ήθελα να μάθω από τους καλεσμένους μας ποιο είναι το μοντέλο που θεωρούν ότι είναι κατάλληλο για την πιστοποίηση. Μιλήσαμε για πιστοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είδαμε τώρα από την κρίση τι κινδύνους ε, επιφέρει αυτό και βεβαίως ε, και τις, ε, τα συγκρουόμενα συμφέροντα, αλλά από την άλλη έχουμε περίπλοκα και πολύ δυσκίνητα συστήματα του δημοσίου τομέα. Τι προτείνετε λοιπόν. Ευχαριστώ. Μαρκο για δεν είναι εδώ. Βερνάρ Μονό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία ανάκαμψης της τυκλοποίησης προκαλεί αντιρρήσεις από πλευράς μας. Μιλήσατε για τα STS και για την αναθεώρηση του CRR. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των νομικών ρυθμίσεων και είναι σε θέση να πετύχουν το στόχο που θέτεται. Η ανάκαμψη της τιτλοποίησης STS θα βοηθήσει υποτίθεται ε, στη χρηματοδότηση, θα ανακάμψει την οικονομία και οι τράπεζες θα βρουν μια καλύτερη δανειοδοτική ικανότητα. Η Ένωση Αγορών Κεφαλαίων λέει ότι θα πρέπει να αποτραπεζοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις για τις μικρομεσαίες. Πώς θα συμμετέχουν λοιπόν οι τράπεζες. Μας λέτε ότι πρέπει να αποφύγουμε τα προηγούμενα λάθη και τις κρίσεις του παρελθόντος μέσω των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών και σωστής αξιολόγησης των κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχει θέμα σε σχέση με το ποσοστό το οποίο μπορεί να κρατά ο εκδότης, το 5%. Ελπίζουμε να μην χαμηλώσει ακόμα περισσότερο. Η έλλειψη ρυθμίσεων για την τυπλοποίηση των συνθετική μορφή είναι σε αντίθεση με αυτό το οποίο επιδιώκεται. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε επίσης τις αλυσιδωτές τυπλοποίησεις. Λέτε ότι θα θέσετε τέλος στις υπερβολές των κριτηρίων που προέρχονται από τις εταιρείες και τους οίκους αξιολόγησης. Πόσο μάλλον που στο τροποποιημένο CRR η εξωτερική ε, αξιολόγηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μιλάτε για απλούστευση, αλλά όταν διαβάζουμε το τροποποιημένο CRR, ο όρος απλούστευση δεν είναι και πολύ συμβατός. Κλείνοντας, πολλοί επαγγελματίες ε, έχουν αμφιβολίες για τις επιπτώσεις ε, του κειμένου για την ανάκαμψη μιας αγοράς που θεωρείται νεκρή. Νομίζω ότι θα πρέπει οι διευκολύνσεις που έχουν γίνει προς τις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δώρο του κυρίου Χιλ προς την χρηματαγορά την Αγγλική, της οποίας ήταν λόμπιστ για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η τυκλοποίηση οδηγεί στην καταστροφή που ζήσαμε ήδη το 8. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας. Thank you. Uh, thank you, Chair. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από χρόνος έχει περάσει θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες βασικές ερωτήσεις. Για την διακράτηση του κινδύνου ήμουν νομίζω σαφής. θεωρούμε πως ε, μια χαμηλότερη ρύθμιση θα ήταν καλύτερη και επαρκής για τα ABCP, ένα περίπλοκο ζήτημα. Στην προηγούμενη έκθεσή μας, εμείς ήμασταν η πρώτη αρχή που ανέπτυξε συγκεκριμένα κριτήρια για την τίτλοποίηση αυτή. Και όταν μάλιστα τα αναπτύξαμε αυτά, είχαν μια συντηρητική στάση για τον αλλαγή της ε, λήξης. Αλλά αντιλαμβανόμαστε πως η συζήτηση αυτή είναι ακόμα ανοιχτή παγκοσμίω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της ε, αγοράς τίτλοποίησης είναι το θέμα της ε, στήριξης ρευστότητας των εκδοτών και βεβαίως ε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο και στηρίζει πάρα πολύ την ε, επιτυχία και την ρευστότητα του προϊόντος αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αποτελεί ένα κίνδυνο για τον ισολογισμό των τραπεζών κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη όσον αφορά την επιστοποίηση από τρίτους εμείς είμαστε επιφυλακτικοί γιατί βεβαίως συμφωνούμε με κάποιες παρατηρήσεις και η από τρίτα μέρη βεβαίως ε, έχει κάποιους κίνδυνους μειώνει τα κίνητρα του εκδότη να διασφαλίσει και να πιστοποιήσει ότι ε, ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Δεν ε, αφαιρεί τα ζητήματα ερμηνείας, οπότε αυτό βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει ρόλος δημοσίων φορέων και βεβαίως υπάρχει και η δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, την οποία θα πρέπει να περιορίσουμε στο βαθμό του δυνατού και να υπάρχει και σοβαρή υποπτία. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια αυτά και την ισορροπία μεταξύ αυτών θεωρούμε πως υπάρχει μια καλή ισορροπία για να υπάρξει και μια αναζωογόνηση της αγοράς. Συμφωνούμε με την άποψη ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα ολιστικά από τη σκοπιά του επενδυτή. Πρέπει να δούμε πώς ζήτηση θα έχει αυτή η τίτλοποίηση, γιατί βεβαίως οι επενδυτές ε, διαλέγουν μεταξύ πολλών προϊόντων, ε, μεταξύ των οποίων και ομόλογα, τα οποία καλύπτονται. Οπότε όταν αναλύουμε τη ζήτηση αυτών των προϊόντων πρέπει να δούμε το ζήτημα συνολικά. Θα σταματήσω εδώ για να αφήσω χρόνο και στους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Έγιναν αρκετές ερωτήσεις για το ποσοστό διακράτησης 20%. Έγιναν κάποια σχόλια με τα οποία συμφωνώ. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί διεθνώς και το είχαμε συζητήσει όταν είχαμε πρώτο ξεκινήσει. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια, κάποιος κανόνας από ακαδημαϊκή σκοπιά ή από κάποια άλλη που μας λέει ότι το 5% δεν λειτουργεί. Οι διπλοποιήσεις ευρωπαϊκές λειτουργήσαν καλά. Και όπως η η μου, αν δεν έχει χαλάσει δεν υπάρχει λόγος να το φτιάχνουμε. Γιατί το μόνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα και το ποσό κεφαλαίου που μπορεί να ε, διατεθεί για δανεισμό. Χωρίς να έχουμε κάποιο ουσιαστικό λόγο. Ε, έγιναν διάφορα σχόλια για το καθεστώς ε, της πιστοποίησης. Να σας πω ότι Μιλάμε για 13 διαφορετικές ε, χώρες. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό να πηγαίνουμε σε 13 ε, διαφορετικές χώρες για να κάνουμε ερμηνεία των κριτηρίων αυτών. Εμείς ε, θέλουμε και ήδη αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχουμε στις τιτλοποιήσεις μας μέσω των όσων καθορίζει η οδηγία ε, περί ενημερωτικών δελτίων. Βεβαίω, αυτά τα οποία μας λένε τράπεζες θεωρούμε ότι είναι γεγονός, δηλαδή ότι αυτό είναι ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, στεγαστικών ή αυτοκινήτων. τώρα, αν κάποιος αμφιβάλλει για τα κριτήριά μας, για το αν έχουμε αρκετή εμπειρία για το χαρτοφυλάκιο δανείων σε μια χώρα. Ε, τι σημαίνει αρκετή εμπειρία. Μπορούμε να πούμε πως θεωρούμε πως ε, αυτό ισχύει και να σας εξηγήσω και γιατί, αλλά τώρα αυτό δεν ξέρω εάν μπορεί να αποτελέσει ε, θέμα αστικής ευθύνης. Γι' αυτό θεωρούμε πως χρειάζεται ακριβώς η βοήθεια τρίτων φορέων πιστοποίησης και θεωρούμε πως η EBA θα έπρεπε να λάβει αυτή τη δουλειά δεδομένη της εμπειρίας της. Για να υπάρχει μια συνεπής ερμηνεία. Υπήρξαν ερωτήσεις για την βάση δεδομένων. Θεωρούμε και είμαστε υπέρ της ε, διαφάνειας ε, των δεδομένων όπως ανέφερα στα σχολιά μου και εγώ και πολλοί άλλοι βάζουμε τα λεφτά μας εκεί πέρα. Δεν λέμε λόγια του αέρα, χρηματοδοτούμε ακριβώς αυτή την βάση δεδομένων. Θέλουμε λοιπόν οι επενδυτές να καταλάβουν τι αγοράζουν από μας. Όχι να τους πουλήσουμε κάτι το οποίο δεν κατανοούν. Τέλος, υπήρξε μια ερώτηση για την ε, ιεραρχία των κεφαλαίων. Είπαμε πως ε, θέλουμε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο η πρόταση του MBA και πληροφορίες ενδιαμέσω. Αυτό είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, όμως είναι ένα μόλις βήμα και φοβάμαι ότι δεν επαρκεί. Γιατί θα πρέπει ακριβώς να δούμε τις κεφαλαιακές ρυθμίσεις που είναι πολύ υψηλές όπως ανέφερε και ο συνάδελφος. Δεν έχουμε βγάλει εκτός τα άσχημα. Έχουν μείνει μόνο τα θετικά και παρέχουμε νομίζω διαφάνεια και δεδομένα ε, αν πληρούμε όλα αυτά τα κριτήρια γιατί ταυτόχρονα ε, τιμωρούμαστε με επιπρόσθετες κεφαλαιακές χρεώσεις ε, που θα καταστήσουν την χρήση της τιτλοποίησης όπως είπε και ο κύριος Φερνάντες θα βοηθήσουν την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής με τον να υπάρχει περισσότερος δανεισμός στην αγορά. Σας ευχαριστώ. κύριος Μέισμερ. Θα εστιαστώ και εγώ στα ερωτήματα περί ABCP. Ένα ερώτημα ήταν τι, πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις γενικότερα. Η αγορά αυτή στην Ευρώπη κυρίως τίτλοποιεί προσδοκόμενα έσοδα, γύρω στο 50% και αυτά πολλούνται απευθείας ε, από τις επιχειρήσεις. Συνήθως ε, οι απαιτήσει αυτές ε, είναι μεταξύ 15 και 50 εκατομμυρίων ευρώ. ευρώ. Δηλαδή, Θα έλεγα από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ήδη επιλέξιμες για αυτή την αγορά, γιατί συχνά είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν έχουν κάποια αξιολόγηση, έχουν απλά μια πρόσβαση σε άλλα εργαλεία των χρηματοχωρών. Οπότε η χρήση αυτής της χρηματοδότησης είναι ένα έξυπνο εργαλείο για αυτές για να έχουν άλλη μια πηγή χρηματοδότησης πέρα από ένα δάνειο τράπεζας τα άλλα μισά, το άλλο μισό των στοιχείων αυτού του προγράμματος είναι δάνεια για αυτοκίνητα και τέτοιες μισθώσεις. Και όπως είπα και στην δήλωσή μου, βλέπουμε πως οι κατασκευαστές ε, μηχανολογικού εξοπλισμού. Έχουν θηγατρικές εταιρείες χρηματοδότησης που προσφέρουν στις ε, μικρές, ε, στους μικρές πελάτες, στους μικρούς πελάτες, με συγχωρείτε, στις μικρές εταιρείες, την δυνατότητα αυτή μέσω του leasing. Οι εταιρείε αυτές leasing χρειάζονται ένα χρηματοδότηση. Ε, ένα χρηματοδότηση αυτή νομίζω είναι ιδεώδης ε, κλάση για τα προϊόντα αυτά. Οπότε, μια μέση επιχείρηση μέσω άμεσης πώλησης των απαιτήσεών της εποφελείται από ένα τέτοιο προϊόν. Ειδικά το θέμα της μίσθωσης με φέρνει σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε πριν, δηλαδή εάν μπορεί μία απέτηση για leasing να είναι επιλέξιμη υπό το καθεστώς αυτό και η πρόταση αυτή λέει πως λόγω των ανησυχιών για την λήξη η μέση ζωή ενός τέτοιου προϊόντος δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος. Έτσι λοιπόν σχεδόν αποκλείονται οι απαιτήσει για μίσθωση γιατί βεβαίω προφανώ διαρκούν περισσότερο από ένα έτο. Οπότε με τον κανονισμό αυτό αποκλείουμε τον κλάδο του leasing από το να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση αυτή